Colleghi, buongiorno, vi invito a prendere posto. Allora, cari colleghi, se non avete obiezioni vi propongo di adottare... συνάδελφοι, αν δεν έχετε αντίρρηση, προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη που έχετε λάβει. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι, ωραία. Να Προτείνω επίση να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδριαση στις 18 και 19 Μαρτίου. Υπάρχουν αντιρρήσει. Εάν όχι, εγκρίνουμε τα πρακτικά. Σημείο 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Καταρχήν μετά από αίτημα του ΕΛΚ, παρέμβαση ενός ε, ειδικού της Ευρωπόλ για τις αρχές του απογεύματος που θα μιλήσει για την παράνομη εμπορία όπλων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διανεμηθεί λοιπόν το πρόγραμμα με την ενημέρωση, με την αλλαγή αυτή. Ε, επίσης σας ανακοινώθηκε από το mail ότι η συνεδρία των συντονιστών που είχε προβλεφθεί αρχικά στις 5.30 το απόγευμα ακυρώθηκε, αναβλήθηκε γιατί δεν υπάρχουν επίγοντα θέματα για μια τέτοια συνεδρίαση. Τελευταία παρατήρηση, αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά μια επιστολή που σας απίφθηνα πριν από κάποιες εβδομάδες προς εσάς, αλλά και που βασικά απευθυνόταν στον πρόεδρο Σούλτσε. Θα θυμάστε πως κάποιες εβδομάδες πριν διάφορες ενώσεις ε, και ιδρύματα κατά της μαφίας, καθώς και συγγενείς θυμάτων της μαφίας και δημοσιογράφοι, ε, απίφθηναν σαφή έκκληση προς αυτή την Επιτροπή, όπου ζητούσαν να κάνουμε κάτι όσον αφορά τον Αντώνιο Δηματέο, ε, τον ε, ειδικό δικαστή κατά της μαφίας ε, του Παλέρμο. Τι έχει συνέβη, τους συμβεί. Τους δύο τελευταίους μήνες στάσανε μια σειρά από ανώνυμες επιστολές με τακτική συχνότητα και εκεί αναφέρεται η ημερομηνία του Μαΐου εντός της οποίας θα δολοφονηθεί από τη μαφία ο εισαγγελέας Ματέο. εντοπίζεται ως ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να ε, είναι ένας από τους ε, ε, δολοφόνους του Ματέου και λέει πως έχει μετανιώσει και ότι δεν θέλει να είναι πλέον μέλος αυτής της δολοφονίας. Έχει δώσει και ένα σωρό πληροφορίες λέγοντας πως τους τελευταίους δύο μήνες ο Ντιματέο, ο οποίος συνοδεύεται από αστυνομία ασφαλείας σε ψηλό επίπεδο στην Ιταλία, έδωσε συγκεκριμένες ενδείξεις, πράγμα που σημαίνει ότι σύμφωνα με τις ερευνητικές αρχές πως ο δικαστής παρακολουθείται για δύο μήνες περίπου και έχουν κάνει πολύ συγκεκριμένε αναφορέ. Αυτό που γράφει είναι πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίο έχει παρακολουθήσει τον Τιματέο όλη αυτή την περίοδο. Επίση, λέει ότι δεν θα πρέπει να παίρνει συγκεκριμένου δρόμου ή στενά δρομάκια. πάντω ε, από εκείνη την ημέρα και μετά συνεχίζουν να φτάνουν άλλες ανώνυμες επιστολές, όπως σας είπαμε πολύ τακτικό ρυθμό, όπου Γίνονται κάποιες αναφορές, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε η, η έκκληση που απευθύνθηκε στην Επιτροπή μας. Ένα από τα τελευταία γράμματα λέει ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα να κάνετε έκκληση στην Επιτροπή κατά της Μαφίας της Ευρώπης. Εμείς έχουμε αποφασίσει ούτως ή άλλως να δολοφονήσουμε τον εισαγγελέα Νίνο Ντιματέο εντός του Μαΐου. Σας ε, καλώ να, δώσετε μεγάλη προσοχή γιατί το ίδιο ακριβώς έγινε το 1992 όταν σκοτώθηκε ο δικαστής Μπορσελίνο και ο δικαστής Φαλκόνε ε, Είχαν σταλεί αυτές οι ανώνυμες επιστολές με συγκεκριμένη περιγραφή των όσων θα γίνονταν και παρόλα αυτά δυστυχώς έγιναν όλα αυτά μετά. Υλοποιήθηκαν. Σημερίζουμε αυτή την έκκληση και μάλιστα την στείλα και στον πρόεδρο Σούλτ. Έχουμε συγκεκριμένη ευθύνη γιατί σε αυτή την έκκληση διάφορες προσωπικότητες του κόσμου της δίωξης της μαφίας στρέφονται σε εμά με την ελπίδα, με βαθιά ελπίδα, ε, λέγοντάς μας δώστε μας μια αναπάντηση τουλάχιστον εσείς, γιατί στην Ιταλία είμαστε χωρίς κυβέρνηση και φαίνεται πως η πολιτική δεν νοιάζεται για τη ζωή και για την τύχη του εισαγγελέα Νίνο Ντιματέ. Εγώ λοιπόν σήμερα θα έρθω σε επαφή με τον ε, πρόεδρο Σούλ να δούμε τι πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε άμεσα. Ε, σήμερα κιόλας ε, θα κάνω ένα σημείωμα προ όλου του συντονιστέ της Επιτροπής μας για να ζητήσω μια επίγουσα ακρόαση ε, ώστε ο εισαγγελέας Ντιματέο να έρθει εδώ και φυσικά θα γίνει και κλεισμένο το θυρόν, δεδομένης τη σημασία των όσων θα μπορούσε να μας πει ο ίδιος ο κ. Ντιματέο. και λόγω όλης αυτής της σειράς ανωνύμων επιστολών που εξακολουθούν να φτάνουν, να καταφθάνουν με συγκεκριμένο ρυθμό. Και σας θυμίζω και υπογραμμίζω ότι οι εισαγγελίες οι οποίοι ερευνούν για αυτά τα θέματα είναι αυτή της εισαγγελίας της καλτενιζέτα οι οποίοι δυστυχώς είπαν πως αυτές οι επιστολές δυστυχώς είναι ε, αληθινές πραγματικές. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, αν συμφωνείτε με αυτή την πρωτοβουλία, θέλετε να πείτε τι πιστεύετε, δεν ξέρω. Παρακαλώ κυρία Μπορσελίνο. Δεν άκουσα εξ αρχής την παρέμβαση, αλλά συμμερίζομαι της, ε, τη μεγάλη ανησυχία διότι είναι κάτι το αισθητό παντού σε σχέση με όλα αυτά, με τα τεκτενόμενα στην Ιταλία. Αυτά τα νέα πέρασαν σε δεύτερο πλάνο λοιπόν εξαιτίας της, ε, της πολιτικής ε, συγκυρίας. Φαίνεται λοιπόν ότι επαναλαμβάνεται η κατάσταση πολιτικής αστάθειας του 1992. Οι ίδιοι οι δικαστές και η εισαγγελία τόνισαν ότι ενυπάρχει αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό θα πρέπει να υπαγρυπνούμε και συμφωνώ ότι ε, θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά σοβαρά υπόψη. Ως προς την ακρόαση, νομίζω ότι οι εισαγγελείς θέλουν να ε, εισακουστούν. Δεν, είναι, δεν πρόκειται μόνο για τον δικαστή Ντιματέο. Πρόκειται και για έναν άλλο δικαστή, το όνομα του οποίου δεν εδόθη, αλλά ξέρουμε ποιος είναι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα γύρω από το οποίο πρέπει να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπορσελίνο, πράγματι αναφέρεστε σε έναν άλλο ε, δικαστή που δουλεύει στην εισαγγελία της Καντανισέτα και μετακινείται μεταξύ Παλέρμο και Καντανισέτα. Το έχουν αποσταλεί πολλά ανώνυμα γράμματα, ότι δηλαδή ε, υπάρχει κίνδυνος να δολοφονηθεί όταν ακριβώς κάνει αυτή τη ε, διαδρομή σε καθημερινή βάση. Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ. Βεβαίω είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα αυτό και ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε. Αναρωτιέμαι, αυτή η Επιτροπή μας τι μπορεί να κάνει. Η απάντηση δυστυχώς είναι τίποτα. Δεν είμαστε εκτελεστική επιτροπή, δεν έχουμε κάποια εξουσία, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε και ακόμα και με το να κάνουμε μια ακρόαση, έστω και κλεισμένων των θυρών, νομίζω ότι απλώς δημιουργούμε προσδοκίες, τις οποίες όμως δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε. Και σε όλη την διάρκεια της εργασίας αυτής της Επιτροπής θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η Επιτροπή δεν είναι Ιταλική Επιτροπή και η Ιταλία έχει προβλήματα και όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν προβλήματα. Ε, συμμερίζομαι απολύτως και πραγματικά σοκάρομαι με αυτά που ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργεί προσδοκίες που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Γιατί οι Ιταλοί πολίτες μετά θα περιμένουν από εμάς να κάνουμε κάτι και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ανησυχούμε, ναι, αλλά έχουμε διαφορετικά εξαιρετική δουλειά να κάνουμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο και δεν θα πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό. Δεν είμαστε Ιταλική Επιτροπή. Ε, Σε σχέση με την εντολή της Επιτροπής δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, ο δικαστής Ντιματέο εργάστηκε επί των θεμάτων που μας απασχολούν, άρα γνωρίζει πολύ καλά την εντολή της Επιτροπής μας, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Η αλληλεγγύη δεν αρκεί πάντα. Όπως είπε και η συνάδελφος Μπορσελίνο, θα πρέπει να τους ακούσουμε, να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει και η Ευρώπη να γνωρίζει, να είναι κοινωνός αυτών των ε, γεγονότων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ως ε, ε, παρατηρητές άλλη μία δολοφονία. Πρόκειται για 12 μήνες, 12 μήνες όπου γίνεται λόγος για τη μαφία στις, ε, στα 27 κράτη-μέλη. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ιταλία, γιατί είδαμε πως η μαφία δυστυχώς έχει τέτοιες διακλαδώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που πρέπει να αντιδράσουμε. Η Επιτροπή Επιτροπή αξιολόγησε πολλά αιτήματα που προήλθαν από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Δηλαδή αξιολογήσαμε τις ε, καταστάσεις, ίσως δεν είναι τόσο σοβαρές σαν τη δική μας, αλλά τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος διακινδυνεύει να σκοτωθεί, δηλαδή να πάει σαν πρόβατο επί σφαγή, δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε μια τέτοια κατάσταση ή να επαναλαμβάνεται στο διηνεκές. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Δεν πιστεύει κανείς ότι η Επιτροπή θα κάνει θαύματα διότι το επίπεδο ασφάλειας ε, έχει ενισχυθεί από τις αρμόδιες αρχές ε, ε, έναντι του δόκτωρα Δηματέου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γνωστοποιηθεί ευρέως αυτή η κατάσταση, γιατί ξέχασα να σας πω και κάτι άλλο. Η Επιτροπή μίλασε, μίλησε και ασχολήθηκε ε, με μία υπόθεση κατά της μαφίας στην Ιταλία και θεωρήσαμε ότι έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μία σαφή ιδέα για το πώς λειτουργεί η μαφία και όχι μόνο στην Ιταλία. Διαφορετικά ε, θα δείξουμε ότι δεν έχουμε κατανοήσει τίποτα από όλους αυτούς τους μήνες ακροάσεων η μαφία έχει καταφέρει να διεισδύσει στα θεσμικά όργανα και στην πολιτική. Εμείς ε, μιλάμε για εκατοντάδες ε, σελίδες, χιλιάδες σελίδες και η ίδια εισαγγελία που ε, παρακολούθησε αυτή τη διαδικασία και έκανε και τις ανακρίσεις σε αυτή την επιτροπή συμμετέχει και ο δόκτωρ Ντιματέο. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο μας απασχόλησε, εκφραστήκαμε και είπαμε ότι θέλουμε να κατανοήσουμε και να ξέρουμε πώς θα διενεργηθεί ή πώς διενεργήθηκε μέχρι τούδε αυτή η δίκη. Βεβαίως ε, για μας είναι όνειδος αυτό, αλλά είναι μια κατάσταση ε, την οποία, στην οποία δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε έτσι, να πούμε εντάξει έχουμε και άλλα να κάνουμε και δεν μπορούμε. Εντάξει, συμπαραστεκόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Δηματία. Η κυρία Ματιέ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη συλλογιστική της Ιταλίας αποκλειστικά βεβαίως. Υπάρχουν δικαστές που δέχονται απειλή για τη ζωή τους. Τώρα δεν έχει σημασία από πού προέρχονταν, είναι Ιταλοί, Βούλγαροι, Ούγγροι και ούτω καθεξής. Θα πρέπει στην Επιτροπή μας να θίξουμε αυτό το θέμα και κλεισμένων των θύρων, αλλά θα ήθελα να ακουστεί και ο Επίτροπος ή Επίτροπος. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει τη μαρτυρία του εν λόγω δικαστή. Αυτό προτείνω. Και να ζητήσουμε και την ε, ε, παρουσία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Ο κύριος Νιούτον Ντάν. Γνωρίζετε την άποψή μου. Είπαμε όχι στην βουλγαρική έρευνα. Δεν την ε, ε, συνεχίσαμε και δεν δώσαμε συνέχεια ούτε και σε, θέματα άλλων εθνικότητων και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να δαπανίσουμε χρόνο εδώ σε αυτή την Επιτροπή που είναι πολύτιμος χρόνος για ένα ιταλικό εσωτερικό θέμα. Είπατε και ίδια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, έπειτα είπατε να τα πούμε στην Ευρώπη τι συμβαίνει, αλλά μετά τα πούμε, κάνουμε και κλεισμένο των θυρών. Άρα δεν θα πούμε τίποτα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Α μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Ήδη έχουμε μείνει πίσω στο πρόγραμμα τη Επιτροπή. Προσπαθούμε να συζητήσουμε τι τροπολογίε. Χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρόνο. Α πούμε, όχι. Α προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Σάλμπρεκτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, ότι όντω χρειαζόμαστε το χρόνο που πρέπει για να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει στην Επιτροπή μα. Έχουμε και την ενδιάμεση έκθεση, έχουμε τα συμπεράσματα τη Επιτροπή μα που πρέπει να το ολοκληρώσουμε και ειλικρινά πρέπει να πω ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο και έχω την αίσθηση ότι και με βάση την ημερήσια διάταξη που έχουμε και όσα έχουμε να διακπεραιώσουμε δεν θα προλάβουμε, δεν θα καταφέρουμε σοβαρά να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε μία έκθεση η οποία θα έχει επαρκή βάση στο Κοινοβούλιο, η οποία να μπορεί να γίνει δεχτή με τα συμπεράσματα που θα προωθηθούν μετά σε νομοθετικές πράξεις. Σωστό είναι βέβαια να ασχοληθούμε με την κατάσταση αυτή, έτσι όπως ε, το κάνουμε εδώ και μισή ώρα. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια την ώρα αυτή για την, να δούμε τις τροπολογίες, ε, γιατί έχουμε και κάποια άλλα θέματα. Εγώ ήρθα για να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες και τις θεωρώ Οπότε μπορώ μόνο να συμφωνήσω με αυτά που λέει ο κύριο Νιούτον Ντάν. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε αυτής της επιτροπή, τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Είναι απολύτως σωστό να πούμε ότι θα στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο στην Ευρώπη, ότι θα το φροντίσουμε με, πολιτικές, με πολιτικά συμπεράσματα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτά τα γεγονότα και ποια είναι η θέση που θα πάρουμε γενικώ, όχι όμω για κάθε ε, μεμονωμένη από ε, περίπτωση που μα απασχολεί. Γενικώ, ποια είναι τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε με του ε, βουλευτέ εδώ και νομίζω ότι είναι και βασική μας, βασικό μα καθήκον. Οπότε α επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι τώρα απαραίτητο να γίνει και αυτό είναι η έκθεση και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να την συζητήσουμε επαρκώ γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικέ οπτικέ για το ποιο θα πρέπει να είναι, ποιο θα πρέπει να είναι ο πυρήνα τη έκθεση, ποια θα πρέπει να είναι τα συμπεράσματα που θα εξαρθούν. Οπότε, αν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτή την έκθεση, εγώ το θεωρώ σωστό. Θα πρέπει να πάρουμε αυτόν τον ε, έξτρα χρόνο. Οπότε ίσω αυτή τη στιγμή α μην δαπανούμε το χρόνο μα σε άλλα θέματα, τα οποία ίσω να μπορέσουμε να κάνουμε. Α συζητήσουμε πρώτα αυτό που έχουμε εδώ πέρα και που είναι το καθήκον μα, που είναι το καθήκον τη Επιτροπή μα. Αυτό μα ζήτησε το Κοινοβούλιο να κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ. Eh, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Έχω την εντύπωση ότι η συμβιβαστική λύση που προτείνει η κυρία Ματιέ θα μπορούσε να μας βρει σύμφωνος. Το θέμα που συνδέεται με την ασφάλεια των εισαγγελέων και των δικαστών, όπου και αν αυτοί εργάζονται, είναι πρόβλημα σίγουρα ευρωπαϊκό, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει νόημα μια επιτροπή κατά του οργανωμένου εγκλήματος με ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση. Πολύ σύντομα λοιπόν, γιατί έχει δίκιο και ο Άλμπερτ που λέει ότι πρέπει να, να συνεχίσουμε και να εξετάσουμε τις τροπολογίες και εκείνες τις συμβιβαστικές. Να πούμε ότι η πρόταση λοιπόν, τη λύση μάλλον της Βερονίκη Μαρτιέ, έχω την εντύπωση ότι είναι σωστή. Θα πρέπει να βρούμε χρόνο και με την Επίτροπο, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση της Σικελίας. Ε, τώρα, αν υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις σε άλλα κρατημέλη, θα ήταν ευκταίο και σε αυτή την περίπτωση να προχωρήσουμε σε ακρόασεις ε, και με άλλους ε, εισαγγελίσει. Ευχαριστώ κυρία Ζόντεργαρντ. Ο κύριος Ζόντεργαρντ, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Αυτό που με σοκάρει περισσότερο σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες που μόλις ακούσαμε είναι ότι οι Ιταλικές αρχές από ό,τι φαίνεται δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν αυτόν τον άνθρωπο παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες απειλές κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς σίγουρα δεν μπορούμε να λύσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ωστόσο, θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί του πολίτες του ε, ακόμα και όταν υπάρχουν εκπεφρασμένες απειλές ε, εκ των προτέρων. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλετε μια επιστολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και να του ζητήσετε να εξεταστεί το θέμα σε ένα άλλο επίπεδο ώστε να ενεργήσουμε και απέναντι στις ιταλικέ αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ματιέ. να πούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε μια συμβιβαστική Μήπως θα μπορούσαμε με την Επίτροπο να μιλήσουμε για την προστασία των δικαστών και των εισαγγελέων γιατί πιστεύω πως σε κάθε κράτος μέλος, σε κάποια κράτη-μέλη έχουν υπάρξει απειλές κατά κάποιων εισαγγελέων. Στη χώρα μου ήδη υπήρξαν απειλές κατά εισαγγελέων που ειδικεύονται στην καταπολέμηση και στη δίωξη της τρομοκρατίας, στην Ιταλία στους εισαγγελείς ε, κατά της μαφίας και, φυσικά, πιθανότατα θα έχουν υπάρξει και σε άλλα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε λοιπόν την Επίτροπο στην Επιτροπή για το έγκλημα, ώστε να μιλήσουμε για αυτό το δύσκολο πρόβλημα και να δούμε αν η Κομισιόν θα μπορούσε κάτι να κάνει, να προβλέψει κάτι, να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση σε αυτό το θέμα. Έτσι θα ξεφύγουμε από το Ιταλικό πρόβλημα. Όντω, γιατί έχουμε την η συνήθεια στην Επιτροπή μα να μην ασχολούμαστε συγκεκριμένα με κράτο μέλο. Αυτό επέλεξαν οι συντονιστέ, όπω είπε και ο Μπιλ, και έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του δικαστικού μηχανισμού. Αυτό προτείνω. Ευχαριστώ. Κυρία Μπορσελίνο, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Ματιό γιατί ακριβώς δεν πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα κρατημέλη και όλος ιδιαίτερος για την Ιταλία, αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό, επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε πολλές χώρες όπου οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι ανακριτές απειλούνται, να κάνουμε όντως μια πιο γενική συζήτηση. Γιατί κιόλας δεν μπορούμε να πούμε πως η Ιταλία δεν προστατεύει τον εισαγγελέα Ντι Οι εισαγγελεί δυστυχώς ειδικά στη συγγελία υπερπροστατεύονται αλλά κάποιες φορές ακόμα και αυτή η προστασία δεν αποδεικνύεται επαρκής απέναντι στην τεράστια ισχύ της μαφίας. Ε, το πρόβλημα λοιπόν του οργανωμένου εγκλήματος είναι ένα πρόβλημα εξαιρετικά διαδεδομένο και είναι δίκαιο να το μιλάμε τόσο όσον υπάρχουν συγκεκριμένες υποθέσεις όσο και όταν μιλάμε γενικότερα. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο και εγώ συμφωνώ. Θα στείλω επιστολή σε όλους τους συντονιστές όπου θα συνοψίζεται η πρόταση της κυρίας Ματιέ και εγώ θα πρέπει να πω σε ταλίδα. δεν νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω για την Ιταλία ε, και να πω ότι δεν μπορούν οι Ιταλικές ε, δυνάμεις να, ε, να προστατεύσουν τον κύριο Ντιματέο. Ταξιδεύει με τρία αυτοκίνητα κάθε φορά τεθωρακισμένα. Το σπίτι του προστατεύεται, αλλά Δυστυχώ, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι η μαφία ακόμα και έτσι μπορεί να ενεργήσει. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όπως προτείνει και η κυρία Ντιματιέ. Ε, και βρίσκω πως είναι καλή η, η πρότασή σας να καλέσουμε και την Επίτροπο και τον Εισαγγελέα. Ξεκινήσουμε με το σημείο 4. Ο εισηγητής κ. Γιακολίνο παρουσίασε το ενδιάμεσο σχέδιο έκθεσής του ακριβώ στην τελευταία μας συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου και μετά από την παρουσίαση του σχεδίου Υποβλήθηκαν από τους διάφορους συναδέλφους 744 τροπολογίες σκιώδεις εισηγητές και οι άλλοι συντάκτες των τροπολογιών έκαναν πολύ πολύ σκληρή δουλειά, εντατική εργασία ώστε να αναλύσουν όλες τις τροπολογίες και να βρουν ε, συμβιβαστικές ε, ώστε να καλύψουν όλες τις ε, δυνατότητες για το τελικό κείμενο. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της συζήτησης, να διαποσαφηνίσουμε τις θέσεις των διαφόρων συντακτών των τροπολογιών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στον κύριο Ιακολίνο για 15 λεπτά για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες και έπειτα 3 λεπτά θα δώσω χρόνο ομιλία σε όλους τους βουλευτές. Φυσικά δίνοντας προτεραιότητα στους συντονιστές όπως προβλέπει ο κανονισμός και έπειτα θα δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Γιακολίνο για να μας απαντήσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας θυμίσω επίσης ότι σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες και τους συντονιστές έχουμε αλλάξει την ε, ημερομηνία ψηφοφορίας που θα είναι η 7η Μαΐου στις 9 το πρωί. Κύριε Γιακολίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως είπατε λίγο πριν, έχουμε 744 τροπολογίες επικοδομητικές σε γενικές γραμμές που προέρχονται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν περιμέναμε την αθρώα αυτή η έλευση τόσων τροπολογιών, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας προσπαθεί να συνεισφέρει και αυτό έγινε μέχρι τις 26 Μαρτίου. Είχαμε μία σειρά συναντήσεων με τους Σκιώδης που ήταν επικοδημητικές πριν από την υποβολή τροπολογιών αλλά και μέσως μετά. Το 1 τρίτον αυτών των τροπολογιών οδήγησαν σε τροπολογίες συμβιβασμού. Φτάσαμε σε 55 συνολικά τροπολογίες συμβιβασμού που διαβιβάστηκαν στις ομάδες. Έχουμε 55 στο σύνολό τους. Εξετάστηκαν από τις πολιτικές ομάδες και εγκρίθηκαν χτες ε, κατά την τελευταία συνάντηση με τους Κιώδης. Σας υπενθυμίζω τα βασικά στοιχεία αυτής της έκθεσης μετά από τις προτάσεις των συναδέλφων. Όλοι γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης, όπως θέλουμε να φτάσουμε σε αυτήν μετά τις τροπολογίες, στην τελική της μορφή δηλαδή. Θέλουμε να καταδικάσουμε κάθε δραστηριότητα της μαφίας στα κράτη-μέλη και τις εκφοβιστικές ενέργειες της μαφίας έτσι ώστε να πρωτοπορήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Μιλάμε Επίσης και για την ε, εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, η οποία να μπορεί να γίνει και σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό της ε, λήψης της απόφασης, μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και στα πλαίσια της συνδρομής ε, αστυνομικών και δικαστικών αρχών και σε τρίτες χώρες. Μιλάμε και για αυτή τη διαδικασία ανακύκλωσης όπως, ε, γίνεται σε όπως ισχύει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτά τα είδαμε στις τροπολογίες συμβιβασμού. Ως προς τη διαφθορά προβλέπεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς και μιλάμε για τη διαφθορά ε, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Επίσης, λάβαμε υπόψη ορισμένες απαιτήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ευάλωτους τομείς που σχετίζονται με τη διαφθορά και ως προς την ανακύκλωση βρώμικου χρήματος θα πρέπει να έχουμε συνεργασία των τραπεζικών αρχών, των συμβολεογράφων και των επιχειρηματιών έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά σε διεθνές επίπεδο. Θέλουμε την ε, συμμετοχή της Eurojust και της Europol, καθώς και του Οργανισμού Υπέρ των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχει ένας, ε, μία αρχή ότι οι επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά και για άλλα σημαντικά εγκλήματα να αποκλειστούν για πέντε ή περισσότερα χρόνια από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε τους έντιμους επιχειρηματίες. Επίσης, μιλήσαμε για την ανιχνευσιμότητα, τη διαδικασία ανιχνευσιμότητας. Ε, ιδιαίτερα προς την παράνομη εμπορία όπλων και των τσιγάρων καθώς και των αλκοολούχων ποτών. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Επίσης, Υπάρχει ένα κέντρο πληροφορικής και πληροφόρησης για τις ε, διεθνείς εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει αυτός ο φορέας οργανισμός που ελέγχει τις ευαίσθητες πληροφορίες και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ανταλλαγή πληροφοριών, μία διαδικασία best practice και συνεργασία, συμφωνίες συνεργασίες με τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι έχει σημασία και το θέμα της κατάρτισης και εκεί προβλέπουμε επικοδομητικό διάλογο με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και την αρρωγή των δικαστικών αρχών και εισαγγελέων. Ως προς την ανακύκλωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι πληροφορίες που λάβαμε πρόσφατα θεωρούν ότι πρόκειται για ε, χίλια δις ευρώ και μιλώ για τις παράνομες δραστηριότητες. Αυτή είναι η προβολή που γίνεται για το 14-20. Και εδώ μιλάμε για την παράνομη, για τη μαύρη οικονομία, η οποία σχετίζεται και με εγκληματικές δραστηριότητες διεθνούς χαρακτήρα. Μιλάμε για παράνομη εμπορία των ναρκωτικών, μεταξύ άλλων, και μιλήσαμε και για διεθνές ε, ή διεθνικό έγκλημα το οποίο θα πρέπει να καταπολεμηθεί για να ε, υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε εγγυητές των δικαιωμάτων της μέσα στα πλαίσια των ε, δυνατοτήτων που υπάρχουν και μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις τρίτες χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε δια... μηχανισμούς διαφάνειας και άρσης της γραφειοκρατίας στη δημόσια διοίκηση. Όσο περισσότερη γραφειοκρατία υπάρχει, εκεί ακριβώς μπορούν να δράσουν, μπορεί να δράσουν οι μηχανισμοί διαφθοράς. Επίσης, το τραπεζικό απόρριτο θα πρέπει να αρθεί διότι πολύ συχνά μπορεί να τροφοδοτήσει το σύστημα ανακύκλωσης βρώμικου χρήματος και είπαμε ότι θα πρέπει οι φορολογικές αρχές να συνεργαστούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αναφερθήκαμε και στην εγγύηση διαφάνειας και πρόληψης και στο, στη διαδικασία πρόσβασης και θεωρήσαμε ότι τα κόμματα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας, του κώδικα δεοντολογίας που θα πρέπει να ισχύει στα πολιτικά κόμματα και πρόσωπα. Μιλήσαμε επίσης για την μη εκλογιμότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη γενικότερα και μιλήσαμε για αναλογικότητα και επικουρικότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την εσωτερική ένομη τάξη των κρατών μελών. Θεωρούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα, η διαφορά και η ανακύκλωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αποφυγής ή πρόληψης ως προς τη διαφθορά, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να ε, διενεργούνται και οι δίκες έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παραγραφής κάποιας δραστηριότητας που να ενέχει στοιχεία διαφθοράς μέσα στα πλαίσια του ποινικού. Μιλήσαμε και για κατασχέσεις. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η μαφία δρά γιατί διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και οικονομικά. Αν λοιπόν άρουμε αυτά τα μέσα, τότε ε, στην ουσία θα συρρυκνωθεί η μαφία. Υπάρχει διαδικασία φυλάκισης και αυστηρής φυλάκισης και κάθυρξης, αλλά και από τη φυλακή ο έγκλειστος μπορεί να δίνει εντολές προς τα έξω. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιπρόσθετο σύστημα όπου στην ουσία να καταπολεμηθεί η ανακύκλωση βρώμικου χρήματος και μέσω μιας τραπεζικής ε, ένωσης για την οποία εργαζόμαστε στεναρά. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πλαισιώσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και θεωρούμε ότι και η διαδικασία κατάσχεσης είναι ύψης της σημασίας για την ανάκτηση πόρων που διαφορετικά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Μέσα στα πλαίσια των ε, συνταγματικών δικαιωμάτων του κατηγορούμενου. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθεί και η διαδικασία κατάσχεση σε όλα τα νομοθετικά συστήματα, ακόμα και για τα παράνομα στοιχήματα. Επίσης, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την καταναγκαστική εργασία και τη δουλεμπορία θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες και αντιμετώπιση με βάση την οδηγία που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και όλους όσους συνεργάστηκαν, η Προεδρία, η Γραμματεία, γιατί πρόκειται για μια δραστηριότητα που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Είχαμε αρχικά 44 τροπολογίες, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε εύκολα. Άρα, πέσαμε στη δουλειά και φτάσαμε σε πολύ καλά αποτελέσματα. Και στην προσεχή συνεδρίαση με τους Χιώδης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σας ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ζήρισε το λόγο ο κύριος Σταβάρης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ νόμιζα ότι πριν θα μιλούσαν οι συντονιστές και γι' αυτό ε, δεν ε, περίμενα μέσω τώρα να παρέμβω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω δύο λόγια. Ε, να πω πώς βλέπω αυτή την ε, διάμεση έκθεση αυτής της Επιτροπής και την ίδια την Επιτροπή. Πιστεύω πως ο ρόλος αυτής της Επιτροπής είναι βασικά πολιτικής φύσης, δηλαδή να υποβάλει συστάσεις για τις δραστηριότητες τις μελλοντικέ της Ένωσης που θα είναι πολύ σημαντικές ε, από την κατάσχεση προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η και ένα σωρό άλλα. Και επιπλέον θεωρώ πως αυτή η έκθεση η ενδιάμεσα πρέπει να είναι πολιτικός ε, πολύ ισχυρή και να λαμβάνει υπόψη πτυχές ε, θεμελιώδους δικαίου, ε, θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικών ελευθεριών και όλα αυτά να διοχετεύονται και μέσα στις πολιτικές. Γιατί αν ήμασταν μέσα στο πλαίσιο μιας νομοθετικής επιτροπής, πιθανότατα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμένε από τις τροπολογίες που αφορούν δικαιώματα, ελευθερίες και εγγυήσεις απερίτευαν, γιατί φυσικά περιλαμβάνονται στις συνθήκες, στα συντάγματα, στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, ούτω ή άλλω οφείλουμε να σεβόμαστε αυτέ τι αρχέ, αλλά καθώ πρόκειται για πολιτικό λόγο, για να δώσουμε πολιτικέ κατευθύνσει, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτέ τι τροπολογίε περιττέ. αντιθέτω μάλιστα. Ε, και αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια των σκιωδών εισηγητών, να εγγυηθούμε ότι αν θεωρούμε πως χρειάζεται να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματο. Γνωρίζουμε πως πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά, να το τονίσουμε όμω αυτό και είναι σημαντικό, όπω λέγαμε ας πούμε για το ξέπλυμα παράνομων προσόδων, φοροδιαφυγή ή επιθετική φοροδιαφυγή που πολύ συχνά ε, συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα ή ακολουθεί τι ίδιε οδού που ακολουθεί το οργανωμένο έγκλημα. Όπως είδαμε πολλές φορές εντός της Επιτροπής και μάλιστα επιβεβαιώθηκε και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Χέρμαν Φαρομπόη, η Ένωση χάνει ένα, τρεις, τρεις ευρώ ετησίως λόγω αυτών των πρακτικών και αυτό αποτελεί τεράστια κοινωνική ζημιά. Και έτσι πρέπει να το παρουσιάσουμε και στην έκθεσή μας ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αλλά μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί μόνο όχι μέσω ενός αγώνα ασφάλειας ώστε να έχουμε όλα τα μέσα, υπηρεσίες, ε, οργανισμούς ε, και αρχές αλλά να γίνει αυτό με όλες τις βάσεις, αρχές, δικαιώματα και εγγύησεις. Γι' αυτό και δεν θέλω να μείνω εκτός αυτής της, της έκθεσης της ενδιάμεσης, γιατί Ήδη βλέπουμε την εντολή της Ευρωπόλ. Όπως ξέρουμε, η Ευρωπόλ είναι ένας οργανισμός συντονισμού των αστυνομικών αρχών ε, των χωρών μας. Εδώ και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είδαμε πολλές φορές ότι η Ευρωπόλ πολύ ελληματικό, ελληματικά αναφέρεται στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή υπολείπεται πολύ όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο και δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια ή μεγαλύτερη εξουσίε εάν δεν υπάρχει και περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος και περισσότερες εγγυήσεις, δικαιώματα, ε, ε εμείς ε, είδαμε 15 συμβαστικές τροπολογίες. Πάλι έχουμε δύο φορές παραπάνω από ό,τι προβλέπαμε. Χρειάζεται όπως έλεγα, όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη για να μην αφήσουμε εκτός ε, κάτι ε, που αφορά τα δικαιώματα της ελευθερίας και της εγγύησης και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά στη συνεδρίαση των σκιωδών ξεκινώντας από απόψε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και τώρα έχει το λόγο η κυρία Ματιέ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους που κατέθεσαν ε, τροπολογίες. 744 τροπολογίες, ειλικρινά δεν περιμέναμε τόση επιτυχία για αυτή την έκθεσή μου, αλλά αυτό φανερώνει πως ε, πολύ ενδιαφέρουν τα θέματα της Επιτροπής μας τους συναδέλφους. Όταν βλέπω πόσο πολύ ασχολήθηκαν οι συνάδελφοι, βέβαια ε, μας χαροποιεί αυτό. Βέβαια είναι πολύ δουλειά για τον εισηγητή, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να εργαστούμε από αυτές τις έκθεση. Δεν μπόρεσα ακόμα να δω τις 55 συμβαστικές τροπολογίες, γιατί με βάση τα όσα μου είπε ο εισηγητής εχθές το βράδυ μόλις τις επεξεργάστηκε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να... Ε, ε, τα δούμε λίγο ψύχρεμα, να δούμε πώς θα δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις ε, συμβιβαστικές, ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, το ξέπλυμα κεφαλαίων χρημάτων, για να ετοιμάσουμε και την τελική έκθεση της Επιτροπής μας. Έχουμε δουλέψει πολύ για αυτά τα θέματα, έχουμε πολύ αφιερώσει χρόνο και θα πρέπει η Ολομέλεια και οι συνάδελφοι που δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν εδώ να το συνειδητοποιήσουν, καθώς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δούνε τι έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτήν την πληγή. Υπάρχουν διάφορες νέες ιδέες για την ενίσχυση της διαφάνειας. Η μίλησε για το τραπεζικό απόρριτο ε, που θα πρέπει να καταργηθεί. Αυτή είναι μια πολύ δυνατή, έντονη ιδέα που δεν θα πρέπει να καταργηθεί, γιατί πρέπει όντως να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έγινε λόγος επίσης για κατάσχεση ε, που είναι στην καρδιά της συζήτηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε γιατί είναι μια ιδέα κλειδί και ο συνάδελφος Ταβάρες μίλησε για την Ευρωπόλ, πρέπει να δοθούν περισσότερα μέσα στην Ευρωπόλ, περισσότερα για την ε, κυβερνοεγκληματικότητα. Τις προάλλες ε, μιλούσα, ήμουνα στην ε, Επιτροπή όταν ο Διευθυντής της Ευρωπόλ μας παρουσίασε την έκθεση και πραγματικά μας προκάλεσε ρίγη όταν δούμε την έκθεση αυτή. Γιατί, σας καλώ όλους να το διαβάσετε, γιατί είναι πολύ συμπληρωματικό όσα κάνουμε εδώ στην Επιτροπή Κρίμα να βλέπουμε και τα νούμερα και να βλέπουμε και τις ε, τάσεις που, ε, στις οποίες έχει καταλήξει η υπηρεσία της Ευρωπόλ. Ε, όπως σας έλεγα, είναι όλα αυτά παραπληρωματικά. 3.600 εγκληματικέ οργανώσεις, τάσεις, ε, φόβοι για την παιδοπορνογραφία, εγκληματικότητα. Πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε για όλα αυτά και να ζητήσουμε περισσότερα μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ελαφρύνουμε την πίεση. Αυτό είναι ο ρόλο τη Επιτροπή μα και ο ρόλο κάθε Ευρωβουλευτή στην Κρήμη και στην ΛΥΜΠΕ για να υπάρξουν περισσότερα χρήματα στην Ευρω... που θα δοθούν στην Ευρωπόλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία λεπτά έχουμε μονάχα, οπότε δεν θα αρχίσω να εξηγώ τις 75 ε, τροπολογίες μου, γιατί θα χρειαστώ δυόμιση δευτερόλεπτα για την κάθε μια. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και σε αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι τα βασικά σημεία. Εδώ μιλούμε για μια έκθεση ε, καταλόγου δράσεων για την Κομισιόν. Τι περιμένουμε εμείς να κάνει η Κομισιόν για να καθοδηγήσει τα κρατημέλη ώστε να αναλάβουν τι κατάλληλε δράσει γιατί αυτά έχουν τη δική του οπτική πιο στενή. Οπότε βασικά πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να κάνει κάποια πράγματα και πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή εικόνα όπω είπαμε και πιο πριν, όχι με μονομένα κρατημέλη. Αυτό που θέλουμε να έχουμε ως αποτέλεσμα είναι να εκπαιδεύσουμε και τους συναδέλφους μας στις διάφορες επιτροπές σε διάφορε ομάδε, γιατί θα πρέπει να μελετήσουν την διάβαση έκθεση και να την ψηφίσουν. Πρέπει λοιπόν και εμεί να εκπαιδεύσουμε του συναδέλφου μα και επίση να πω ότι το κόστο του οργανωμένου εγκλήματο είναι τεράστιο. Η Βερονίκ ε, αναφέρθηκε στην έκθεση για την Europol. Μιλούμε δηλαδή για εκατομμύρια θέσει εργασία χαμένε, δισεκατομμύρια χαμένων, χαμένων φόρων, ένα καρκίνωμα που πραγματικά κατατρώει την κοινωνία μας. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε αυτό που έχουμε ε, ε, βρει εμείς σε ό,τι αφορά την έλλειψη συνεργασίας από τις, ε, από τις ακροάσεις μας, έλλειψη συνεργασίας και έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Δεν σου δίνω στοιχεία γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Αυτό όμως είναι αστείο γιατί όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Μιλούμε για 60 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο και πολλοί από αυτούς προστατεύονται από το δικό μου το κράτο. Επίση, ε, έχει πει και ο συνάδελφο ε, Θεόδωρο, που δεν είναι εδώ τώρα, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη διαφθορά. Παντού υπάρχει η διαφθορά και η απάντηση στη διαφθορά είναι η διαφάνεια. Όσο περισσότερο ξέρουμε το τι κάνει ο καθένα, τόσο πιο εύκολο είναι να είμαστε διαφανεί. Όλοι, ένας πρωθυπουργό πριν από 100 χρόνια είχε πει ότι όλη η εξουσία διαφθείρει, αλλά η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απολύτως τους πάντες. Οπότε μιλούμε για διαφθορά που υπάρχει όχι μόνο σε χαμηλά στρώματα, αλλά στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, σε επίπεδα πρωθυπουργών, προέδρων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε όλα τα επίπεδα διαφανείς. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ε, καμιά αστυνομική δύναμη ε, δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα. Το πλεονέκτημα των εγκληματιών είναι ότι αυτοί μπορούν πάρα πολύ εύκολα να περάσουν τα σύνορα. Και επίση κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Europol. Ελπίζω ότι μετά από την επιστροφή των, από τις ΕΠΑ, τη ε, προσωπία μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε το πράσινο φω, ώστε να μπορεί η Europol να γίνει κάτι σαν το FBI ώστε να έχει και αστυνομικέ εποπτικέ εξουσίε. Είναι λοιπόν αυτό ένα καρκίνωμα το οποίο κατατρώει την κοινωνία μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις, ε, τους συναδέλφους μας να μελετήσουν την ενδιάμεση έκθεση γιατί πραγματικά είναι τεράστια ευθύνη που φέρουμε. Ευχαριστώ. Albrecht. Albrecht. συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό ακριβώς που μόλις ε, είπε ο συνάδελφος Νιούτον Ντάν, αλλά και η κυρία Ματιού. Ε, όντως έχουμε τεράστια ευθύνη, πολύ ψηλή ευθύνη για αυτή την έκθεση. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σωστή δουλειά, πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε όλες τις διαφορετικές οπτικές και βεβαίως Υπάρχουν ε, κάποιοι που ανησυχούν ε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων κανόνων. Εδώ κινούμεθα σε έναν τομέα που είναι πολύ ευαίσθητος ε, για τα κρατημέλη. Μιλούμε για ποινικό δίκαιο, μιλούμε για διαδικασίες που απορρέουν από το ποινικό δίκαιο. Τώρα μιλούμε για δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών, ποινικών. Σε αυτό το τομέα λοιπόν πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι αρχές του κράτους δικαίου αλλά και οι συνταγματικές αρχές θα πρέπει να συγχωνευτούν, θα πρέπει να συνδυαστούν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι διαφορετικές νομικές κουλτούρες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και να τις ε, ε, καταγράψουμε. Αν απλώς προσπαθήσουμε χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα κράτους δικαίου και συγκεκριμένες θεμελιώδεις αρχές μέσα στην έκθεσή μας, θα χάσουμε την υποστήριξη πολλών από το Κοινοβούλιο και βεβαίω θα χάσουμε και την εμπιστοσύνη των κρατών μελών. Γιατί αυτό δεν το θέλουμε, γιατί η έκθεση μας πολιτικό πώ είναι σωστή. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Ακριβώς για το τομέα της ε, φορολογική απάτης, του ξεπλήματο μαύρου χρήματος, διαστδιαφθόρας. Βεβαίω υπάρχουν και άλλοι τομείς, το οργανωμένο έγκλημα, το εμπορίο ανθρώπων. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά για να έχουμε την πολιτική στήριξη που θέλουμε, για να μην μπούμε απλώ ότι στο τέλο θα έχουμε μια έκθεση την οποία θα θέλουν πολλοί να αγνοήσουν ακριβώ επειδή κάποια σημεία, κάποια ουσιώδη σημεία δεν περιλαμβάνονται. Θα πρέπει να το αποφύγουμε λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή η έκθεση να, είναι, ε, να έχει το σωστό κέντρο βάρους, να, να δείχνει προς το μέλλον και κυρίως θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Η κυρία Ματιό μίλησε για τη Europol, για τη χρηματοδότηση της Europol. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, γιατί ε, μιλούμε και για τις κοινέ ε, επιχειρησιακές ομάδες αυτό και από τη δική μας την πλευρά θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μήνυμα ότι η καθημερινή συνεργασία των ερευνητών θέλουμε να προωθηθεί. Ο κύριος Νιούτον Ταν επίσης ε, μίλησε γι' αυτό. Είπε για την εμπιστοσύνη των αστυνομικών μεταξύ τους ε, για να δουλέψουν μαζί, να δουλέψουν από κοινού, για να κάνουν μια έρευνα, ή για να κάνουν, ξεκινήσουν μια ποινική διαδικασία. Αυτό πρέπει να προωθήσουμε. Και αυτό πρέπει να, για αυτό, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κοινέ βάσει. Γιατί η εμπιστοσύνη χρειάζεται μια κοινή νομική βάση, κοινού κανόνε. Και ε, θεωρώ ότι σε πολλέ τροπολογίε ε, φαίνεται ότι φοβούνται πολύ ότι δημιουργούμε έτσι ένα, ένα, μια, μια, ένα κενό ας πούμε, μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να, να, να συνεργαστεί αλλά κατά τα λοιπά ε, δεν θα υπάρχει συνεργασία. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε, το είπε και ο συνάδελφος Ταβάρες, ε, κοινέ αρχές, κοινά πρότυπα για τα βασικά δικαιώματα, για την προσέγγιση των δεδομένων, για διαδικασίες, γιατί κάνουμε και τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι βασικές προϋποθέσεις για μια καλύτερη συνεργασία, την οποία βεβαίω επιθυμούμε όλοι. Οπότε, αν δεν τα καταφέρουμε μέσα από την έκθεση να θέσουμε τις βασικές αρχές και να τις προωθήσουμε επιθετικά, δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ να επιτύχουμε την επιθυμία μας για καλύτερη συνεργασία. Και γι' αυτό σας κάνω έκκληση. Οι διαφορετικές οπτικές γωνίες θα πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση και από αυτούς τους ευρωβουλευτές που ε, δεν ασχολούνται καθημερινά ίσως ε, με τη μαφία ή με συγκεκριμένες υποθέσεις ή με οργανωμένο έγκλημα κτλ. Και μπορεί να έχουν και μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά το δικό του το νομικό σύστημα αντιμετώπιση όλων αυτών των ε, θεμάτων. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ μας και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε με όλες τις ομάδες να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Γιατί ε, αν εδώ από την Ειδική Επιτροπή βγει μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο η οποία θα υποστηριχθεί μόνο από τους μισούς ή έστω λίγο πάνω από τους μισούς, ε, τότε προφανώς δεν, είχαμε κανένα, δεν, δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξη. και δεν θα μπορούμε να κάνουμε και τίποτα πρακτικά, δεν θα μπορούμε δηλαδή να αναλάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Οπότε όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, βεβαίω και στον εισηγητή Μιλό και στους Σκιώδης, ας βρούμε από κοινού λύσει έτσι ώστε να υπάρξει ευρεία πλειοψηφία και σε τούτη την Επιτροπή, να καταγραφούν όλες οι απόψει και μετά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτέ και τις υπόλοιπες επιτροπές να τους πείσουμε ότι τα βήματα που έχουμε προτείνει είναι επαρκή. Ευχαριστώ. Grazie adesso. Ευχαριστώ. Ε, ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πραγματικά πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Τρία πράγματα θέλω να πω. για την έκθεση αυτή μιλούμε για το πόσο βαθιά μπορεί να μπει κανείς στο πρόβλημα. Γνωρίζουμε βεβαίω όλοι ο καθένας από τις δικές μας χώρες όταν γίνεται ένα ε, έγκλημα, όταν διαπράττεται ένα έγκλημα ε, όλοι ε, θέλουν, όλοι οι πολιτικοί ζητούν περισσότερες αστυνομικέ δυνάμεις, περισσότερες διεκτικές αρχές κτλ. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς. αν δεν ε, μπούμε στη ρίζα του, δεν φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, ε, τότε δυστυχώς αυτά που βλέπουμε σήμερα θα επαναλαμβάνονται. Κάποια σημεία τώρα, ε, τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και είναι νομίζω σημαντικά σε σχέση με τη συνολική συζήτηση που κάνουμε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Ας πούμε οι ανισότητες μας σε μια κοινωνία οι οποίε αποτελούν ε, τον κινητήριο μοχλό για τέτοιε εγκληματικέ ε, πράξεις. Ε, δημοκρατία, έλλειψη δημοκρατίας, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε εγκληματικέ πράξει, αλλά βεβαίω το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο το οργανωμένο έγκλημα, απτείται πολλών τομέων. Πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι αιτίες και αυτές ε, πρέπει να τις ε, φωτίσουμε. Ε, είναι επίσης σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αστυνομικές δυνάμεις να συνεργάζονται. Βεβαίως, είμαστε όλοι της άποψης ότι η εγκληματικότητα προφανώς ξεπερνάει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μιλούμε για την Κίνα, για την Λατινική Αμερική, για τη Ρωσία. Η εγκληματικότητα κινείται παντού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνουμε εδώ, αυτό που προτείνουμε όταν μιλούμε για αστυνομική συνεργασία, είναι να ε, προτείνεται μια αστυνομική συνεργασία η οποία να μπορεί να λειτουργήσει και εκτό των δικών μα συνόρων. Και να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει μάλλον η ε, συνεργασία και μεταξύ αρχών ε, διαφορετικών χωρών. Αλλιώς θα είναι δύσκολο ε, να συνεργαστούμε εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας εντός. Επίσης σημαντικό είναι να κινητοποιήσουμε και την ε, κοινωνία των πολιτών. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Όταν κάποιος έχει μόνο αστυνόμους οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν με τους ε, πολίτες, δεν μπορεί να, να, αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Ε, οι περισσότερες ε, περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια ήταν άνθρωποι που υποχρεώνονταν να εργαστούν σε κάποιες επιχειρήσεις, εξαναγκάζονταν γυναίκες σε πορνεία. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε υπάρχουν ισχυρά συνδικάτα, ας πούμε, με δημοκρατικά δικαιώματα που μπορούν να παρέμβουν. Έχουμε, κάνει κάποιες, ε, έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες, οι οποίες ακριβώς αφορούν αυτά τα σημεία και θέλουμε να συμπεριληφθούν στο, στην έκθεση του εισηγητή. Βεβαίω, όταν θα έχουμε εξετάσει όλο το α, τμήμα αυτό, προφανώ θα συμμετάχουμε και περαιτέρω στην διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα έλεγε ο Ρουι πριν, ότι δεν είναι νομοθετική έκθεση και κυρίως οι στόχοι της είναι πολιτικής φύσης και πρέπει να είναι φιλόδοξη για αυτό το λόγο γιατί αυτή η Επιτροπή δημιουργήθηκε μετά από μια σημαντική όθηση που φέρνει στην Ευρώπη ένα θέμα το οποίο μέχρι στιγμή έμεινε κάπως στην άκρη και δεν είχε αποσαφινιστεί. Αυτή την ε, σύγχυση ε, εξακολουθώ να τη τονίζω. Το να χρησιμοποιούμε, να λέμε ακόμα μαφία και κλιματικότητα ε, τύπου μαφίας δείχνει ότι αρνούμεθα ότι το οργανωμένο έγκλημα τύπου μαφίας υπάρχει και είναι διαφορετικό από το οργανωμένο έγκλημα όπως αυτό το λέμε. Θα πρέπει καταρχήν λοιπόν να καταλάβουμε ότι ισχύει αυτό. Μιλάμε και για οργανωμένο έγκλημα τύπου μαφίας. Δεν είναι ταυτόσιμη, ούτε αντίστοιχη αυτή η δύο Είναι διαφορετικού τύπου εγκλήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, εδώ σίγουρα δεν μιλάμε για συγκεκριμένες μαφίες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες. Δυστυχώς είναι σαφές πως οι Ιταλικές μαφίες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουν μεγάλη σημασία γιατί έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Και άρα σιγά σιγά έχουμε φτιάξει και τα κατάλληλα μέσα. Ε, συχνά λοιπόν γίνεται λόγος για την Ιταλία. Όχι γιατί θέλουμε να μεταφέρουμε στην Ιταλία, να το περιορίσουμε το πρόβλημα στην Ιταλία, αλλά μόνο και μόνο γιατί ε, έχει μεγαλύτερη σήμαση και δυστυχώς και επειδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα πράγματα και έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα. Και εγώ θεωρώ λοιπόν ότι όταν γίνονται λόγος για τέτοια επιχειρήματα, όχι λόγω της προσωπικής μου ιστορίας, δεν είναι σίγουρα χάσιμο χρόνο ε, το να ασχοληθούμε με μια υπόθεση που εμπίπτει αυτή, στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής. Είναι η Επιτροπή μας που αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα, ορίζεται κάπως περιοριστικά ε, ορισμένες φορές ως Επιτροπή κατά της μαφίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Εφόσον είναι συγκεκριμένη αυτή η Επιτροπή, είναι σαφές πως θα πρέπει να ασχοληθεί με όλα όσα την αφορούν. Και σίγουρα δεν είναι χάσιμο χρόνο το να ασχολούμαστε με το να βρούμε μέσα για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε όλα αυτά τα εγκλήματα. Αυτό είναι ο στόχος αυτής της Επιτροπής. Πέρα από αυτό θέλω να πω ότι το γεγονός ότι υποβλήθηκαν 747 τροπολογίες με εντυπωσίασε βέβαια γιατί και λόγω το πώς είχαν γίνει οι προηγούμενες συζητήσεις αλλά και με ανακούφιση γιατί δεδομένη της λιγοστής συμμετοχής που εν γέννη υπάρχει στις συνεδριάσεις μας οι 740 τροπολογίες σημαίνει πως ένα σωρό συνάδελφοι διάβασαν με προσοχή την έκθεση και βρήκαν ενδιαφέρον και θέλησαν να υπογραμμίσουν τα πράγματα τεράστια δουλειά, γιατί έχει γίνει και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν σημαντικό. Σίγουρα μπορεί να τελειοποιηθεί, γιατί όλο και κάτι μπορεί να μας ξεφύγει, αλλά μπορούμε να το καλύψουμε και να το επανεισάγουμε. Και πιστεύω λοιπόν πως αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να είναι φιλόδοξη, γιατί πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα, μάλλον πρέπει να κάνει πολλά σημαντικά βήματα μπροστά σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμή και όσα έχουν μέχρι τώρα ε, ληφθεί υπόψη. Για να γίνει αυτό νομίζω πως χρειάζεται συνεργασία όλων πραγματικά και ότι ακόμα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, κυρίως να ορίσουμε συγκεκριμένα για ποιο πράγμα μιλάμε. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Ε, συμμερίζομαι απόλυτα την παρέμβασή σας και τα όσα διευκρινίσατε αρχίζοντας και όσα είπε ο κύριος Σταβάρες. Εγώ προσωπικά ε, ευχαριστώ την, τον κύριο Γιακολίνο για την εργασία του και μένα με εντυπωσίασε που είδα τόσες τροπολογίες και λόγω του γεγονότος ότι οι συνεδριάσεις μας δεν είναι τόσο ε, ωστόσο δείχνει πως υπάρχει προσοχή σε σχέση με, τα όσα, με τις εργασίες μας που έχουν καλύψει ένα σωρό θέματα. και όπως σας είπα και για μένα ήταν ε, προσβλητικό αυτό, όχι μόνο λόγω της προσωπικής μου ιστορίας, της δικής μου και της κυρίας Μπορσελίνου, αλλά ενώπιον συγκεκριμένων προβλημάτων που είναι ευρωπαϊκά προβλήματα. Διότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, δεν είναι ένα πρόβλημα μιας χώρας, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί διαφορετικά δεν μιλάμε για κράτη με λί. Και εγώ θεωρώ λοιπόν πως ήταν πολύ σοβαρό, αλλά σίγουρα Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα αθέλητο λάθος το να μιλήσει κανείς για χάσιμο χρόνο. Ε, καλή την πίστη έγινε αυτό από πλευράς κάποιου συναδέλφου. Και συμφωνώ πως υπάρχει και πολιτική ευθύνη καταρχήν από πλευράς της Επιτροπής μας που πρέπει να είναι φιλόδοξη και γιατί όχι. Ακριβώ για να μην αφήσει τίποτα την ελεύθερη μετάφραση, ερμηνεία. Μέρα με τη μέρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε το πεδίο της αβεβαιότητας και της αμφιβολίας. Καλούμεθα να παρουσιάσουμε μια εργασία όσο γίνεται πιο φιλόδοξη. Έχουμε τη δυνατότητα από πολιτικής πλευράς και μη νομοθετικής βέβαια να δώσουμε μια, ένα περαιτέρω input Εφόσον δεν έχουμε αντιμετωπίσει για τους λόγους που εσύ υπογράμμισες την παρουσία τη συγκεκριμένη των οργανωμένων ε, ε, εγκληματιών τύπου μαφίας, ακριβώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, δυνατότητα αυτή που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε και τη διαφθορά, αν χρειάζονται συγκεκριμένα στάνταρ διαφάνεια, σε διαφάνεια που χρειάζεται καταρχήν από πλευρά των πολιτικών. Και άρα σε αυτό εμείς πρέπει να είμαστε όχι μόνο διαφανείς αλλά και ευέλικτοι στο να πάρουμε πληροφορίες, ε, να μάθουμε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Να δώσουμε, δηλαδή, κάποια από τα πρώτα νούμερα που θα μας ζητηθούν. Δηλαδή, όταν ε, δρούν οι οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις ε, ε, αυτό επηρεάζει και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, Όλη αυτή η πλημμύρα από πλημμυρίδα εγκλημάτων που μέχρι στιγμής έχουμε υπογραμμίσει Πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας που να μην κρύβεται πίσω από εύκολες ε, δικαιολογίες όπως εμείς όποτε δεν έχουμε αρμοδιότητα. Και πάνω απ' όλα έχουμε πολιτική ευθύνη και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιακολίνο για να δώσει τη δική του άποψη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα προφανώς με ανανεωμένο ενδιαφέρον τα όσα είπατε και αυτά που είπε η κυρία Μπορσελίνο, ότι πρέπει δηλαδή να βρούμε πολιτική συμφωνία σε υψηλό επίπεδο, ώστε αυτή η έκθεση να είναι μια καλή έκθεση. Δεν μπορούμε μετά από ένα χρόνο ακροάσει, επαφές... ερωτήσεις... να μην φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές και χρήσιμο κυρίως αποτέλεσμα χρήσιμο για τις αστυνομικές αρχές, για τους εισαγγελείς, τους ανακριτές και για τα κράτη-μέλη και για την Κομισιόν που θα πρέπει να έχει Ε, με στόχο να θεσπίσουμε κοινέ νομικές προδιαγραφέ, να εγγυηθούμε προστασία των ε, μετανοημένων, των μαρτύρων, ε, των, των καταγγελόντων και όλων όσων εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις και γι' αυτό και θεωρώ πως είναι σημαντικό, όπως και είπαν και οι συνάδελφοι, αυτό το έργο που κάναμε, ορισμένοι υπέβαλαν απαιτήσει να φτάσουμε δηλαδή στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια με μεγάλη υποστήριξη. Η απόδειξη είναι οι 55 συμβαστικές τροπολογίες που έχουν μέχρι τώρα υποβληθεί, αλλά και η κοινή μας βούληση όλων των βουλευτών του Προεδρείου μας, των συμβούλων μας, να βρούμε δίκαιες και λογικές συμβιβαστικές λύσεις που θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις απαιτήσει κάθε ομάδας. Κανένας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Ε, πρέπει να εγγυηθούμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ταυτόχρονα αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί όριο ή περιορισμό στην άσκηση της δράσης από πλευράς των αρχών τάξης και της ε, εισαγγελίας. Δεν μιλάμε τώρα για κοινό έγκλημα, μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Οργανωμένο με επιστημονικό τρόπο, με μεγάλες δεξιότητες επιχειρηματικές, επιστημονική οργάνωση που μπορεί να κινηθεί χρονικά και διεθνώς. Πρέπει να αυξήσουμε δηλαδή το επίπεδο προσοχής, αλλά κυρίως να είμαστε συγκεκριμένοι και συσπηρωμένοι όσον αφορά τους στόχους μας. Θέλουμε να εργαστούμε λοιπόν εντατικά πάνω σε όλα αυτά. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν αλλά και εκείνους ε, που δεν παρενέβησαν και που θέλησαν απλά να δείξουν την ευαισθησία τους σε σχέση με μια κρίσιμη φάση 7 Μαΐου. Ψηφίζονται οι συμβαστικές τροπολογίες. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε μια άλλη επαφή. Αύριο ε, θα υπάρχουν δυνατότητες για να μπορέσουμε να έχουμε πιστικές παρατηρήσεις. Κυρίως υπάρχει μια κοινή προσπάθεια υπεύθυνη ε, να μπορέσουν δηλαδή καινούρια ε, θεσμικά, ε, θεσμικά όργανα ε, καινοτόμα να δώσουν μια νόθεση. Γι' αυτό προσπαθούμε και εργαζόμαστε εντατικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο για τις απαντήσεις σας και για τις ευκρινήσεις σας. Να θυμίσω πως σίγουρα, σήμερα στις 5.30 έχουμε μια άλλη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε συσπηρωμένη την ομάδα και να δώσουμε μια έκθεση με την οποία θα συμφωνούν όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστούμε κύριε Γιακόλινο και τώρα να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο επιχείρημα ανακύκλωση χρήματος και φοροδιαφυγής στα κράτη-μέλη και συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τον Μάικλ Ντέβαλτ από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Γερμανικής Αστυνομίας που θα εξηγήσει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης και της φοροδιαφυγής από την άποψη της Γερμανίας. Έπειτα θα ακούσουμε τον Ντομαγκό Ιμπαριέτο που είναι, από την ε, διευθυντή, ε, που είναι δημοσιογράφος έρευνας και θα μιλήσει για τη φοροδιαφυγή στις χώρες ένταξης όπως η Κροατία. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Ούγκαρ που είναι καθηγητής ε, του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης για την δημόσια οικονομία και θα δώσει μια ανάλυση για την φοροδιαφυγή και η χρόνοι είναι πάντα ίδιοι. Έχουμε ο κάθε ομιλητής 15 λεπτά για να μας εκθέσει την ε, εισήγησή του και μετά θα αρχίσουμε τη συζήτηση με τρία λεπτά για κάθε βουλευτή. Okay. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, καταρχάς σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ ενώπιν της Επιτροπής σας θα σας ε, μιλήσω για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος ε, μαύρου χρήματος. Θα σας πω ποια είναι η άποψη της γερμανικής ε, πλευράς. Θα σας αναφέρω κάποια βασικά σημεία. Αρχικά θα μιλήσω για το γενικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος στη Γερμανία θα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχουν 40 ε, ε, συστάσεις της ε, ειδική ομάδας για την χρηματοοικονομική δράση. Υπάρχει το, η ομάδα Egmont, υπάρχουν οι διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως σχετικές αποφάσεις. Εγώ είμαι ο επικεφαλής της σχετικής μονάδας στην Γερμανία. Ε, ασχολούμαστε πάρα πολύ με την ομάδα Egmont που ορίζει ε, παγκοσμίω ε, ποιοτικά πρότυπα και όσοι πληρούν αυτά τα πρότυπα γίνονται μέλη της ομάδας Egmont και βεβαίως συνεχίζουν την βελτίωση των κανόνων τους για να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη Γερμανία συγκεκριμένα υπάρχει ο ποινικό κώδικας, παράγραφος 261 για την ποινικοποίηση ε, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και βεβαίως υπάρχει και η σχετική πράξη για, την, για το ξέπλυμα χρήματος όπου ορίζει τα βασικά, ε, τις βασικές προϋποθέσεις ε, κυρίως για την σχετική μονάδα FIU της Γερμανίας. Πολύ σημαντικό είναι, και αυτό θα το πω αρχικά στην παρουσίασή μου, ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ε, ουσιαστικά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν ε, για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος. Ε, γιατί έτσι όπως η συγκέντρωση, έτσι όπως θα σας την παρουσιάσω και στην παρουσίασή μου, ορίζεται κυρίως στην ειδική ομάδα χρηματοοικονομικών δράση, δράσης για το Πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή, πώς εμπλουτίζουμε τα πρότυπα που υπάρχουν ε, για να ξεκινήσουν οι ερευνητικέ διαδικασίες, ε, να μπορούν να δουλέψουν οι διοκτικές αρχές. Βεβαίως υπάρχει και άλλη μία μεγάλη συγκεκριμένη προσέγγιση για όσους θεωρούμε ότι είναι ολοκληρωμένα ή μπορούν να εμπέσουν στην ολοκληρωμένη ε, χρηματοοικονομική έρευνα, δηλαδή στρατηγικές πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε, επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες ε, προέρχονται από τις ε, αρχές ασφαλείας. Πάμε τώρα πίσω στο πρώτο τμήμα για, τις, ε, για τα καθήκοντα που έχει η ομάδα FIU στην Γερμανία. Ε, εδώ ε, αναφέρεται, όλα αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 10 του ποινικού κώδικα. Συνοπτικά αυτά είναι τα καθήκοντά μας, τα βλέπετε. Και βεβαίως αυτά προβλέπονται και από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Ότι δηλαδή έχουμε τους α, υπόπτους, Βεβαίω εδώ έχει γίνει μια ε, διευκρίνηση, δεν μιλούμε ε, για ενδείξεις, ε, αλλά για δήλωση υποψιών. Δεν υπάρχει δηλαδή κατόφλι για τους υπόχρεου να διαβιβάσουν τέτοιες πληροφορίε στην Γερμανία. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα κλασικά καθήκοντα όπω τα βλέπετε, να αναλαμβάνουμε τις διάφορε αυτέ δηλώσει, να τα αναλύουμε και ό,τι θεωρούμε ότι είναι σχετικό και μπορεί να βοηθήσει τι διοκτικέ αρχέ να το προωθούμε. Να το στέλνουμε δηλαδή σε αυτές τις ειδικέ μονάδες που ασχολούνται με τα, θέματα αυτά. με τα θέματα αυτά. Αναλύουμε λοιπόν και λαμβάνουμε, αναλύουμε και διαβιβάζουμε τις ε, σχετικές πληροφορίες. Βλέπετε ότι έχουμε και, άλλες, ε, και άλλα καθήκοντα, δημοσιεύουμε τις ε, εκθέσεις, ενημερώνουμε τους εμπλεκόμενους για τρόπους λειτουργίας που έχουμε, για διάφορες τυπολογίες, λειτουργούμε και, συνεργαζόμαστε μάλλον και με άλλες ομάδες FIU. Αυτά, τουλάχιστον ε, για τα α, καθηκοντά μας, τα υπόλοιπα βεβαίω μπορείτε να τα βρείτε όπως σας είπα στην παράγραφο 10 του ποινικού κώδικα. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση. Από την ε, αρχή της αντιμετώπισης α, ε, της, του ξεπλήματος, από το δηλαδή που ποινικοποιήθηκε το ξέπλυμα, έχει, έχουμε μια σταθερή αύξηση των περιπτώσεων. Η, ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν το 2011, περίπου 13.000 τέτοιες δηλώσεις. Για το 2012 δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη ο αριθμός, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 13.000 για το, 2012 και αν δούμε το, την τάση για το 2013, αν υπολογίσουμε για το, συνολικά το 2013, σίγουρα θα περάσουμε και το όριο του 2012. Για την δημοσίευση των τελευταίων αυτών στατιστικών στοιχείων διαπιστώσαμε και πραγματικά ήταν οδυνηρό ότι στα ΜΜΕ ε, μετά από αυτά τα, μετά τη δημοσίευση αυτών των δεδομένων γινόταν λόγος ότι το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία αυξάνεται. μιλώ ε, ενώπιον, ε, ενώπιον εμπειρογνώμων, αλλά ε, ε, συγχωρήστε με που το λέω. Δυστυχώς ε, μιλούμε και για ε, ε, διαρροή χρημάτων. Προφανώς όσο περισσότερες λεπτομέρειες λαμβάνει κανείς, τόσο περισσότερες υποθέσεις θεωρητικά υπάρχουν. Αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση στη Γερμανία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του, του ξεπλήματος έχει βελτιωθεί όταν υπάρχουν όλο και περισσότεροι ε, αξιωματούχοι στου ε, δρόμους για να κάνουν ακριβώς ε, επιτόπου ελέγχους, προφανώς αυξάνεται ο αριθμός των υποθέσεων που καταγράφουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται το πρόβλημα, σημαίνει ότι το παρακολουθούμε πολύ περισσότερο και καταγράφουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, για την κατανομή των διαφόρων δηλώσεων, των διαφόρων εκθέσεων. Η πλειοψηφία των ε, εκθέσεων αυτών έρχονται από τον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Περίπου 90% ή πάνω από 90% ίσως ε, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Περίπου 90%. Έχουμε 935 από τα ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έχουμε περίπου 6-7-8% ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι λίγο παρόμοια τα, τα αριθμητικά μας στοιχεία με, τους με τις υπόλοιπες χώρες. υπάρχουν και, οι άλλες, και τα άλλα μέρη, τελευταία σειρά, ε, δηλαδή όχι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εκεί βεβαίως χρειάζονται και άλλες, και άλλες πληροφορίες. Ε, βεβαίως το πρώτο βήμα που, που γίνεται είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο βήμα είναι όλα αυτά να αναλυθούν και να αναλυθούν οι δράσεις που πρέπει έτσι ώστε σε αυτό το τομέα να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Ασχολούμαστε λοιπόν πολύ εντατικά. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα συνέλθει ένας, μια συντονιστική ομάδα από όλες τις εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνε για τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε εδώ να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση, να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για να δουν πώς μπορούν να διχειριστούν αυτόν τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Σύντομα, για κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε κάθε χρόνο στις διάφορες εκθέσεις που δημοσιεύουμε. Τα πιο ισχυρά, τα πιο σημαντικά θα σας αναφέρω. Από τις, όλα τα υπόλοιπα βέβαια μπορείτε να τα βρείτε στην ε, ε, ιστοσελίδα μας. Για τις εθνικότητες ε, των ατόμων που έχουν καταγραφεί, βλέπετε εδώ, βεβαίως αναφέρονται οι περισσότεροι, Γι' αυτό και το λέω μάλλον αυτό γιατί ε, παρατηρούμε πάντα ότι τα στατιστικά στοιχεία ε, διαβάζονται ε, πάρα πολύ γρήγορα και δεν σκεφτόμαστε πάρα πολύ το τι ακριβώς σημαίνουν. Δύο πράγματα να πω εδώ. Αυτά είναι εισαγωγικά στατιστικά. Αναφέρεται μόνο τι λαμβάνουμε από τις διάφορες εκθέσεις ό,τι αφορά την, τις προφορίες για την, για την εθνικότητα αυτού του ατόμου. Δεν περιλαμβάνω δηλαδή καμία, άλλο, καμία άλλη πληροφορία για την περαιτέρω διαδικασία. Και επίση, ε, ε, για παράδειγμα, τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε για την Τουρκία, Τούρκου ε, υπηκόου. Θα μπορούσε κανείς να προβληματιστεί. Αλλά αν, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η τουρκική κοινότητα στην η Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλη με πολίτες που έχουν την τουρκική υπηκότητα ή είχαν την τουρκική υπηκότητα. Η κοινότητα λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, επομένω δεν είναι περίεργο που οι Τούρκοι υπήκοοι ε, βρίσκονται σε αρκετά ψηλή θέση εδώ στον πίνακά μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία ε, ε, είναι σαφές το τι ακριβώς σημαίνουν και τι ακριβώς πρέπει να διαβάσουμε πίσω από τα ψυχρά νούμερα. Τώρα, βλέπουμε εδώ ε, αιτήματα που έχουν αποσταλεί στην FIU Γερμανίας. Τα περισσότερα από την Γερμανία, από αστυνομικέ αρχέ γερμανικέ δηλαδή, που θέλουν πληροφορίε ή που θέλουν να συγκρίνουν πληροφορίε με άλλε μονάδε FIU. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Μετά έρχονται αιτήματα από άλλε χώρε. Αυτό που δεν έχουμε εδώ, γιατί ε, ευχαρίστως συγκρίνουμε βέβαια στα δεδομένα μας με άλλες χώρες και βλέπουμε ποιος είναι πιο πάνω, ποιο είναι πιο κάτω, πώς ε, λειτουργεί το πράγμα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε ότι εμείς ε, στη Γερμανία είμαστε αστυνομικοί FIU και λαμβάνουμε πάρα, πολύ, πάρα πολλά αιτήματα που αφορούν ε, αιτήματα που πρέπει να σταλούν προς την Europol ή προς, την, άλλες αστυνομικέ μονάδες. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν διαβάζουμε τέτοια στατιστικά στοιχεία. Τώρα, σε ποιους τομείς, με ποιους τομείς ασχολούμαστε. Δεν θα σας εκπλήξουν εδώ βεβαίω τα στατιστικά στοιχεία, γιατί όσα στατιστικά έχω δει εγώ είναι παρόμοια. Η απάτη είναι συνήθως στην πρώτη θέση, έτσι και στη Γερμανία, 52% περίπου. Α, ναι, αναφέρω το στατιστικό αυτό στοιχείο γιατί εδώ μιλούμε για ε, ε, συνεργασία και με τις φορολογικές αρχές. 2% των δηλώσεων που λαμβάνουμε και αναλύουμε εφόσον έχουν θεωρηθεί σχετικά, διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές για περαιτέρω επεξεργασία. Μετά, από την ανάποδη αν το δούμε, το 2012 πήραμε πάνω από 300 εκθέσεις, πληροφορίες από τις φορολογικές αρχές. σύμφωνα και με, τον, ε, με το τμήμα 31B του φορολογικού κώδικα που επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να στέλνουν αυτές από την πλευρά τους πληροφορίες ε, σε εμά. Μάλιστα δεν επιτρέπεται απλώς, ε, είναι υποχρεωμένες να στέλνουν τις πληροφορίες σε εμά. Σε εμάς. Ειδικά όταν έχουν πληροφορίες για ξέπλυμα μαύρο χρήματος, το οποίο εμπίπτηκε στο, στην παράγραφο 61 του ποινικού μας κώδικα. Αυτά από μένα λοιπόν σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε το ξέπλυμα μαύρο χρήματος στη Γερμανία σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει το λόγο ο Γκόγκ. Μάργκετικ, ο οποίος προέρχεται από την Κροατία, είναι δημοσιογράφος και θα μας ε, μιλήσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροαποφυγή. Ε, έχετε και εσείς 15 λεπτά. Gentlemen, members of the European Parliament. Καλημέρα σας, ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα σας μιλήσω για την περίπτωση της Κροατίας, η οποία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την περίπτωση Χίπο Άλπε Adria όχι μόνο στην Κροατία, αλλά και στα Βαλκάνια και στην Αυστρία. Ε, επειδή είμαι ερευνητής, δημοσιογράφος ερευνητής, ε, θα σας μιλήσω για το σκάνδαλο ΧΥΠΟ, το οποίο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε που ε, άρχισαν οι δραστηριότητες στην Κροατία η θηγατρική στη Κλάγκενφουρτ διέθετε 244 ε, δις 550.000. Στη συνέχεια η Χίπο Κλάγκενφουρτ είχε και μία θηγατρική στο Ζάγκρεπ με 1 δις 581 εκατομμύρια 991.000 ε, κροατικών also bought another Croatian subsidiary uh, uh, called uh, Slavonska Banka Osijek. Και αυτό που μας ενδιέφερε ήταν και η Σλαβόνσκα Μπάνκα η οποία διέθετε 998 ε, δις, 713 εκατομμύρια κροατικά ε, κούνας. Αυτό που με ενδιέφερε εμένα για... είναι να δω από πού προερχόταν αυτό το κεφάλαιο. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην Hippo Άντρια Μπάνκ στην ε, Klagenfurt, η οποία διέθετε και άλλες θηγατρικές και παραρτήματα στα Βαλκάνια. Άρα, από πού προερχόταν ε, αυτά, προέρχονταν αυτά τα χρήματα. Ξέραμε ότι αρχικά ε, υπήρχαν πολλές, ε, ε, πολλά, χρήματα που είχαν διατεθεί στα παρακλάδια στις θυγατρικές και δεν ξέραμε από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Και μέσα στα πλαίσια της ανιχνευσιμότητας ε, είδα ότι υπήρχε ένας ειδικό ε, φάκελος στην Κροατία στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό αφορούσε δραστηριότητα από το 1999 μέχρι το 2001 στην Αυστρία ιδιαίτερα, όπου είδαμε ότι στην Χίπο, στον όμιλο Χίπο Άλπε η υπήρχε και ε, ε, ε, διενεργήθηκε μία έρευνα από την Κροατία και δύο ερευνητές απολύθηκαν ακριβώς επειδή υπήρχε, υπήρχε νομικό υπόβαθρο να συνεχίσει η έρευνα. Αλλά δεν θέλαν να υπακούσουν στα πολιτικά, στις πολιτικές προσταγές για να σταματήσουν αυτή την έρευνα γιατί επρόκειτο για χρήματα τα οποία προέρχονταν από κυβερνητικές πηγές και είχαν υπεξαιρεθεί από το δημόσιο προϋπολογισμό. Από την 14 η μου έρευνα έμαθα ότι τα χρήματα προέρχονταν από κυβερνητικές δημόσιες πηγές από τον ε, δημόσιο τομέα και από την παραοικονομία ως προς το δημόσιο τομέα από που ε, προερχόταν από την ιδιωτικοποίηση. Άρα όλα τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να προέρχονταν από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης κατά τη δεκαετία του 90 δεν έφτασαν στο, στους δημόσιους λογαριασμούς αλλά μεταβιβάστηκαν σε μυστικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που ελέγχονταν από την κυβέρνηση και από το ε, κόμμα της κυβέρνησης. Πρόκειτο για ε, υψηλούς αξιωματικούς της Κροατίας. Και μετά είχαμε και τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά ταμεία, τα χρήματα των οποίων πήγαν σε μυστικούς λογαριασμούς και ελέγχονταν από την Hippo Alpe Adria Bank. και τα χρήματα αυτά δεν πήγανε στους συνταξιούχους γιατί υπεξερεύτηκαν αυτά τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μετά είχαμε το Ταμείο Άμυνας και Ανάπτυξης το οποίο ελεγχόταν από κυβερνητικούς αξιωματούχους και τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν από ε, εμβάσματα, καλύφθηκαν από εμβάσματα ε, για την άμυνα κατά τη δεκαετία του 90 και προέρχονταν από το εξωτερικό από μετανάστες ε, επίσης και τα χρήματα αυτά βρέθηκαν στο εξωτερικό, σε μυστικούς λογαριασμούς. Πάντα τη Χίπο Άλπε Άντρια Μπάνκ με βάση την Klagenfurt. Επίση είχαμε τις αποταμιεύσεις των πολιτών. Κατά τη δεκαετία του 90 οι αποταμιεύσεις των πολιτών εξαφανίστηκαν και η επίσημη εξήγηση από το Ζάγκρεπ ήταν ότι αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν ε, στο Βελιγράδι και μετά δεν έγινε ε, εκ νέου μεταφορά στο Ζάγκρεπ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα, διότι αυτά τα χρήματα ε, μεταβιβάστηκαν σε μυστικούς ε, λογαριασμούς στο εξωτερικό και έφτασαν στην Κλάγκενφουρτ, στην Χίπο Άλπε Άντρια Μπάνκ. Επίσης είχαμε δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποίησαν μυστικούς λογαριασμούς του κυβερνώντος κόμματος και μετέφεραν αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για δις ε, κούνας από τις δημόσιες επιχειρήσεις σε μυστικούς ε, λογαριασμούς στο εξωτερικό, οι οποίοι ελέγχονταν ε, βεβαίως, επρόκειτο για ένα δίκτυο, ένα μαύρο δίκτυο λογαριασμών. Επίσης είχαμε και την ιδιωτικοποίηση στον τομέα της ε, στέγης και στέγασης, όπου μέσα στα πλαίσια της ε, ιδιωτικοποίησης μπορούσαν να αγοράσουν τα σπίτια τους οι πολίτες και φτάσαν αυτά τα χρήματα σε μυστικούς ε, λογαριασμούς στο εξωτερικό. Αυτό αφορούσε και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των τραπεζών. Τα χρήματα φτάσαν στους μυστικούς αυτούς λογαριασμούς και βεβαίως Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από φορολόγηση των ε, πολιτών και η, Zagreb, η τράπεζα Zagreb Batska Bank μετέφερε αυτά τα χρήματα στην χιπο Alpe Adria Bank από το Zagreb στο Klagenfurt Επίσης, τα χρήματα αυτά της ε, Κροατίας που μεταφέρθηκαν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να βοηθήσουν τους εκεί πολίτες, υπεξαιρέθηκαν αυτά τα χρήματα και βρέθηκαν σε μυστικούς λογαριασμούς. Ίσως ξέρετε και το σκάνδαλο της ε, ε, Σεργοβάτσκα Μπάνκ. Επίσης είχαμε και τα συγκεκριμένα ταμεία, μαύρα ταμεία, τα οποία προήλθαν από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες όπου συμμετείχε και η κυβέρνηση. Από το πετρέλαιο, από ναρκωτικά, από ε, παράνομη εμπορία τσιγάρων και από ε, τοξικά, ε, τοξικά απόβλητα τα οποία ε, έτυχαν αυτής της ε, δραστηριότητας παράνομης εμπορίας. Από ε, τις παράνομες δραστηριότητες ξέρετε δηλαδή την περίπτωση ίσως της Zagreb Bank. Εδώ βλέπετε τα, το δίκτυο των τραπεζών που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία ξεπλήματος και στα Βαλκάνια, όχι μόνο στην Κροατία. Κατά τη διάρκεια του 1990, ξέρετε την εμπόλεμη κατάσταση που επικράτησε στα Βαλκάνια και μέσα στα πλαίσια αυτής της αλληλεξόντισης και ο Τουσμαν και ο Μιλόσεβης είχαν κοινέ δραστηριότητες και να σας πω και για την δραστηριότητα στη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο τη Σλαβόνσκα Μπάνκ. Και το βρώμικο χρήμα μεταφέρθηκε σε αυτούς τους μυστικούς λογαριασμούς. Και όταν άρχισε αυτή η διερευνητική δραστηριότητα, ε, αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην Χίπο Άλπε Άντρια Μπάνκ. Πώς ε, το κατέφεραν, κατάφεραν. Είχαν ενδιάμεσους, εντολοδόχους, ε, αξιωματούχους, ε, ανθρώπους του υποκόσμου και των τραπεζών, καθώς και επιχειρηματίες. Δηλαδή, όποιος είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κροατία ή τραπεζικές δραστηριότητες, καθώς και τα εγκληματικά δίκτυα, συμμετείχαν σε αυτή τη ε, διαδικασία ξεπλήματος από επιχειρηματίες και από τον, ακόμα και τον πρώην ε, Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταδικαστεί. Βλέπετε εδώ επίσης ε, το δίκτυο διοικητικών επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου Τραπεζών, και βλέπετε όλους τους επικεφαλείς ε, δικτύων του υποκόσμου που συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος και την επίσημη ελίτ. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να μην έχει συμμετάσχει σε αυτές τις εγκληματικές ε, δραστηριότητες, είτε μέσα στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης, είτε ε, μέσα στα πλαίσια παράνομων δραστηριοτήτων και εμπορίας πετρελαίου, τσιγάρων και ούτω καθεξής. Τι έκανε λοιπόν ε, το κράτος, μετέφερε αυτά τα ε, χρήματα σε λογαριασμούς, μυστικούς λογαριασμούς με βάση συγκεκριμένους εντολοδόχους, και η βασική δραστηριότητα ήταν της Hippo Alpe Adria Bank, η οποία έκανε επενδύσεις, συγκεκριμένες επενδύσεις μέσα στα πλαίσια των ε, ιδιωτικοποιήσεων, τουριστικών ε, δραστηριοτήτων και ούτω καθεξής. Τι έκαναν. Ε, έπαιρναν τα χρήματα και τα ε, μετέφεραν στην Hippo Alpe Adria Bank στην Klagenfurt Εάν σας ενδιαφέρει μπορώ να σας δώσω και τα ε, στοιχεία υποστήριξης. Ε, πρόκειτο για ε, καταθέσεις από τη θηγατρική, από την μητρική με συγχωρείτε, στις ε, θυγατρικές και επρόκειτο για μυστικούς λογαριασμούς σε τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αγορά ομολόγων και μετοχών και ούτω καθεξής. Δηλαδή κάθε μεγιστάνας ε, της Κροατίας σχετίζεται με αυτό το σκάνδαλο της ε, Hippo Alpe Adria Bank και έγινε μεγιστάνας με βάση αυτή τη δραστηριότητα. Επίσης υπήρχαν και καταθέσεις στο Λίχτενστάιν, στα Βαλκάνια στο Λίχτενστάιν είχαμε 55 ε, τέτοιες φορείς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια λοιπόν του 90 χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι μαύροι λογαριασμοί οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτό τον όμιλο. Από το 95 μέχρι το 99 τι οι πόροι ε, πήγαν σε μυστικούς λογαριασμούς στην Χίπο Άλπε Άντρια της Κλάγκενφουρτ και ήταν ο βασικός φορέας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Επίσης, ο Όμιλος Χίπο ήταν ένας από τους βασικούς τραπεζικούς εταίρους ε, της κυβέρνησης και οι περισσότεροι υψηλοί αξιωματούχοι εργάστηκαν γι' αυτό, συνεργάστηκαν με τον όμιλο της Χιποάλπε Άντρια Group και αυτό αφορά και τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καταδικαστεί. Επίσης και πρώην μέλη του Κοινοβουλίου έχουν καταδικαστεί μέσα αυτές, στα πλαίσια αυτών των παρανόμων δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η Μπριγκίτε Ούγκερ που είναι λέκτορ στο, Πανεπιστήμιο της Ιουτρέχτης. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα, επειδή γεννήθηκα Αυστριακή και τρέχει στις φλέβες μου κροατικό αίμα. Διδάσκω ε, στην Ολλανδία και είμαι και διευθυντή ενός Γερμανικού Ερευνητικού Ινστιτούτου. Αισθάνομαι πολύ Ευρωπαία ε, και με έχουν πολύ συγκινήσει οι ομιλίες των προηγούμενων ομιλητών. Θέλω να σας μιλήσω για τη τελευταία ανάλυση όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ε, πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια έκθεση προς την DG Home ε, για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής περί ξεπλύματος χρήματος στις 27 χώρες. Η έκθεση αυτή δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί και αυτή είναι η μονάδα μου που βλέπετε εκεί και κάθεται. Ε, να σας πω μόνο κάποια πρώτα σημεία και τα υπόλοιπα θα δημοσιευθούν ε, πολύ σύντομα, προσεχώς. Ε, βασικά λέμε ότι υπάρχει αυτή η απειλή που είναι πολύ διαφορετική στις διάφορες χώρες. αναλύσαμε πώς εφάρμοσαν τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς εκτέλεσαν την νομοθεσία αυτή, τα όσα μας είπε ο προηγούμενος ομιλητής για τη Γερμανία, ο κ. Ντέβαλτ. Επίσης, πώς έγιναν όλα αυτά μέσω της δημόσιας ε, ε, ε, δίωξης, και πώς τελικά έχουν, έχει γίνει, είχε μάλλον ασκηθεί η ποινή στις διάφορες χώρες. Να δούμε τώρα αν η φοροδιαφυγή ε, είναι η ίδια. Ε, η απειλή που βρήκαμε είναι κάτι είναι κάτι σημαντικό από όγκο. Δηλαδή, αν τα χρήματα από τα ναρκωτικά και τα χρήματα από διαφθορά πήγαιναν του κόσμου πήγαιναν σε ευρωπαϊκές χώρες, πού θα πήγαιναν. Δεν σημαίνει πως πραγματικά πηγαίνουν εκεί αυτά τα χρήματα, αλλά ποιες χώρες είναι πιο ελκυστικές. Εδώ βλέπουμε τις κόκκινες χώρες που βλέπετε εδώ και δείτε τη γεωγραφία. Είναι σαφώς οι δυτικές, οι πλούσιες χώρες που είναι ελκυστικές για τους πλήστες. Η Κύπρος θα δείτε πως δεν είναι σε αυτόν τον κατάλογο. This is in percent of GDP. Επόμενη σπίνακα ε, είναι καλύτερο. Εδώ είναι στατιστικέ, ο βαθμό των οποίων προσελκύει σε σχέση με το ε, ε, πώ απειλούνται οι χώρε και είναι μικρότερε χώρες και εκεί βλέπουμε ότι είναι μικρότερε χώρε και εκεί Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό νησάκι το οποίο κινδυνεύει. Εστονία, το, Λετωνία επίση το ίδιο και αντιμετωπίζουν μεγάλο όγκο σε σχέση με το μέγεθός τους. Το ξέπημα χρήματος λοιπόν σε όγκο είναι οι μεγαλύτερες χώρες. Ο μεγαλύτερος πλήστης ε, βρώμικου χρήματος είναι η ΙΠΑ, αλλά ποτέ δεν ακούμε να μιλάνε για, την, για, αυτήν, για αυτές μάλλον. Μια γενική παρατήρηση. Είναι πρόσφατο το θέμα. Το 1986 έγινε η πρώτη σχετική νομοθεσία στις ΕΠΑ και προηγούμενα δεν υπήρχε. Όχι ότι δεν προσπαθούσαν οι χώρε να βγάλουν κρυφά χρήματα, αλλά δεν είχε οριστεί εν πάση περιπτώσει. Διεθνεί προδιαγραφέ το 1989 από τι G7, ε, τι πλουσιότερε χώρε του κόσμου και διαδόθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Μέχρι στιγμή μόνο τέσσερι χώρε δεν καλύπτονται με κάποιο τρόπο από τι προδιαγραφέ ξεπλήματο χρήματο. Όλε οι υπόλοιπε έχουν γίνει δεκτέ. Είτε είναι μέλη του IMTF, είτε του περιφερειακού περιφερειακών σωμάτων του FTF έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Επίσης έχει επεκταθεί από τον αλκάπόνη στην Αλκάιντα έχει πάει. Αρχικά ήταν τα χρήματα των ναρκωτικών, αλλά τελικά έχουμε διαφθόρα, χρηματοδότηση τρομοκρατία, φοροδιαφύγη, ένα σωρό πράγματα καλύπτονται. Και μέχρι και την ε, εξάπλωση των όπλων και έπειτα υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ε, φορέων αλλά και αντίσταση και προβλήματα συμμόρφωσης όταν διευρύνονται οι προδιαγραφές και διαδίδονται τόσο γρήγορα. Για σας δώσω ένα παράδειγμα, οι δικηγόροι σε πολλές ε, χώρες ανησυχούν για την ιδιωτική ζωή και τα νομικά προνόμια. Όταν δηλαδή έρχεται κάποιος πρέπει κανείς να τον αναφέρει στον κύριο Ντίβαλντ το θέμα είναι έχουμε το νομικό προνόμιο, έχουμε δυνατότητα στην ιδιωτική σφαίρα, στο απόρριτο. Αυτά τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα στην Ευρώπη και δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν. Και έπειτα, ε, για να είναι νόμιμη όλη αυτή η δίωξη, θα πρέπει να είναι πιο ορατή. Ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, συλλογή φόρων, μπορεί να είναι μια ευκαιρία ώστε να είναι μια επιτυχία αυτής της πολιτικής που αγγίζει συμφέροντα πολλών πολλών ανθρώπων. Οι μαύρες λίστες, ε, έτσι όπως δηλαδή διανύμε η η ε, ομάδα δράσης ε, αυτή τη διαδικασία είπε δηλαδή ότι αν δεν ε, συμμορφωθείς θα μπει σε μαύρη λίστα και κανείς δεν θα συνεργάζεται μαζί σου. Αυτή η μαύρη λίστα του FATF θα δείτε ότι άδειασε πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπετε τη μαύρη λίστα του 2006 και έφυγε από την αγορά μια νέα μαύρη λίστα άρχισε να ισχύει το 2009 με περισσότερες χώρες ε, που δεν αντιστέκονται στην, ε, στα, στα σχήματα και στις προδιαγραφές. Εδώ έχουμε δύο χώρες στη μαύρη λίστα. Την, η μία είναι η, μαύρη, είναι η, νότια, η Βόρεια Κορέα και ε, η Τουρκία περιλαμβάνεται σε αυτές τις χώρες που είναι και μέλος του FMTF. Έτσι που οι χώρες αναγκάζονται να κάνουν μια προσπάθεια για να βγουν από το καταλόγιο Γερμανία που επικρίθηκε ότι δεν υπήρχαν αρκετές εκθέσεις αύξησε τις εκθέσεις της αυτές. Ασκείται πίεση που δεν προέρχεται από την οδηγία, αλλά από το FATF και από τις ε, κυρώσεις της μαύρης λίστας. Όταν αναλύσαμε τις 27 χώρες δεν ήταν σαφές κατά πόσο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, ε, στόχο είχε να καταπολεμηθεί η εμπορία ναρκωτικών, της τρομοκρατίας ή η φοροδιαφυγή. Και τα κράτη-μέλη πολλές φορές διαφορετικά ερμηνεύουν τις πολιτικές αυτές. Όταν δούμε την, το πλούτο κάθε χώρας, και Σαφώς θα δούμε πως η καταπολέμηση των ναρκωτικών βασικά αφορά τις χώρες όπου υπάρχει χαμηλότερο κατακεφαλή, ενώ η φοροδιαφαγή είναι η μέρημνα των πιο πλούσιων χωρών. Και μετά έχουμε και τις μπλε οικονομίες, τις, τις ε, πιο κατα... συμπιεσμένες θα λέγαμε. Οπότε η φοροδιαφυγή είναι μέλημα περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Ο ΣΑ επίσης ξεκίνησε με ένα κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Εδώ όπως θα βλέπετε δεν είναι ευρωπαϊκός ε, χάρτης. Πολύ συχνά τίνουμε να βάζουμε την Ευρώπη στο μέση. Εδώ όμως είναι στα αριστερά η Ευρώπη γιατί είναι αυστραλι... αυστραλέζικος ο χάρτης τούτος. Έχουμε λοιπόν το Λιχτεστάιν, το Isle of Man, Μονακό, Ανδόρα, τα βλέπετε στα αριστερά του χάρτη, αλλά ο ΣΑ σαφώς έχει αναγράψει εδώ τις μικρές χώρες, ενώ προηγούμενες οι κατάλογοι έδειχναν πολλές μεγάλες χώρες ως παραδείσους, φορολογικούς παραδείσους. Η Κύπρος δεν είναι σε αυτόν τον κατάλογο πλέον. Γιατί λοιπόν τα φορολογικά έσοδα και η φοροδιαφυγή είναι τόσο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης ο κόσμος, οι χώρες πρέπει να εξοικονομήσουν χρήματα, πρέπει να περιοριστούν οι κρατικές δαπάνες, η κόκκινη γραμμή και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι ε, τα φορολογικά έσοδα μειώνονται Γι' αυτό και η φοροδιαφυγή αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ε, οι μετρήσει λοιπόν τη φοροδιαφυγή δείχνουν ότι η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη αυξάνεται. Εδώ έχω βάλει έξι χώρε, πέντε μάλλον, όπου έχω κάνει εκτιμήσει. Η φοροδιαφυγή λοιπόν αυξάνεται σε όλε αυτέ τι ευρωπαϊκέ χώρε τελευταία, κυρίω μετά από την έναρξη τη οικονομική κρίση. Και κατά με το πρόβλημα ήταν τι είναι φορολογικό έγκλημα, τι είναι φοροδιαφυγή και τι είναι φοροαποφυγή και σε τι θα πρέπει να εστιάσουμε. Με βάση τη νέα πρόταση της οδηγίας που ίσως θα έχετε μελετήσει ή θα μελετήσετε, ε, το θέμα είναι ότι πως δεν περιλαμβάνεται ως εδώ το έγκλημα το φορολογικό, δεν λέει φόρο διαφυγή. Εγώ αρχικά δεν ήμουν ευχαριστημένη που δεν αναφερόταν, αλλά σε λίγο θα σας δείξω κάτι. Όταν ε, διέρευσε το offshore, ε, ε, ήταν κατέστη σαφές ότι πολλές εταιρείες όπως τη Starbucks, στην πιο ακριβή χώρα ας πούμε που δεν έχει καφέ, την Ελβετία, δεν κάνουν φορά διαφυγή, δηλαδή, δεν κάνουν κάτι το παράνομο, κάνουν φόρο αποφυγή και το Βρετανικό Κοινοβούλιο σωστά το καταδίκωσε ως ανήθικη συμπεριφορά και αυτό είχε αντίκτυπο γιατί όταν αγοράζω πλέον ε, καφέ Starbucks ε, ε, το σκέφτομαι πριν Επίσης το ότι διώκονται διάφορες προσωπικότητες γνωστές ε, οδηγεί στο να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρους στις πολιτισμένες κοινωνίες και ότι πρόκειται για ένα έγκλημα, διότι στερείς από το δημόσιο τομέα τα πράγματα που έχει να κάνει για μια κοινωνική Ευρώπη. Για, κατ' το πρόβλημα είναι η φοροδιαφυγή, η φοροαπάτη και η φοροαποφυγή η φοροδιαφυγή θα ήταν, ένα, ε, θα ήταν έγκλημα για τις χώρες όπου μπορώ να διαβάσω και να μελετήσω την, τον ποινικό κώδικα. Διεπίστωσα πως η απάτη είναι έγκλημα στη Γερμανία, την Αυστρία, αλλά μόνο για τις επιχειρήσεις και τις εγκληματικέ οργανώσεις. Δηλαδή η ιδιωτική ε, φοροδιαφυγή δεν θεωρείται έγκλημα για διαφορετικά, στις, στις, στις κάτω χώρες η φοροαποφυγή, η υποφοροδιαφυγή είναι ίσονο σημασία ε, παρανομία. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τι είναι φοροδιαφυγή, είναι ένα φορολογικό έγκλημα, έγκλημα θα, θα το ορίσουμε. Η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα σε κάθε χώρα, αυτό δεν είναι σαφές. Ας πούμε, αν αυτός ο περίφημος ε, γερμανός ποδοσφαιριστής ε, φοροδιαφεύγει, θα θεωρήσουμε ότι κάνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή θα θεωρηθεί ότι κάνει μόνο φοροδιαφύγη. Η νέα οδηγία λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε γιατί η φοροδιαφυγή μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διάφορες χώρες η φορολογική απάτη. Η Κύπρος τώρα. Εγώ δεν κατάλαβα καθόλου τη συζήτηση για την Κύπρο, γιατί έλεγε ότι η Κύπρος έχει ξεπλύνει ε, βρώμικα ε, ρωσικά χρήματα από φοροαπάτες. Για μένα αυτό σήμαινε ε, σύγχυση μεταξύ τριών διαφορετικών πραγμάτων. Καταρχήν έχουμε τις τράπεζες, 7% ε, ε, ε, του ΑΕΠ, 700% του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή 7 φορές μεγαλύτερο από όλη τη χώρα και για οι τράπεζες μεγάλωσαν τόσο πολύ που πολλές από αυτές τις τράπεζες είναι τράπεζες που δεν μπορούν να δανείσουν χρήματα στις επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι η βασική τους δουλειά αυτή. Το τραπεζικό τομέα είναι πρόβλημα ο ίδιο. Σε αυτό οφείλεται η οικονομική κρίση, ήταν το πρόβλημα τη Ιρλανδία, τη Ισλανδία και τη Κύπρου. Και λέει ότι λόγω των, της φοροδιαφυγής και της φυγή ε, φυγής κεφαλαίων των Ρώσων ολιγαρχών που φυσικά γιατί δεν ήθελαν να βάλουν τα λεφτά τους στη Ρωσία, αυτό είναι πρόβλημα για τον κύριο Πούτιν. Δεν είναι δικό μας. Και το τρίτο, ότι είναι λέει ξέπλυμα χρήματο, αυτό με, πραγματικά με μπέρδεψε, γιατί ξέπλυμα χρήματο στην Κύπρο στη δική μας ταξινόμηση βρίσκεται στα μέσα, είναι μέσα στο μέσο όρο. Την ίδια ποιότητα ε, έχουμε όπως σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο. Η Κύπρος δηλαδή δεν είναι καλύτερη χειρότερη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οπότε η σύγχυση ανάμεσα σε αυτά τα, χρήμα, αυτά τα τρία, δηλαδή ότι τα ρωσικά χρήματα ξεπλένονται μέσω των τραπεζών, δεν το κατάλαβα, δεν κατάλαβα γιατί ε, μπερδεύτηκαν όλα αυτά, αλλά νομίζω πως έγινε μια πιο ηθική συζήτηση και όχι μια ε, ξεκάθαρη συζήτηση για την κατάσταση της Κύπρου, πράγμα που νομίζω δεν τάξιζε αυτή η χώρα. Συμπεράσματα. Το φορολογικό έγκλημα είναι μια χαμένη ευκαιρία για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή μέσω συγκεκριμένων νόμων για το ξέπλυμα του χρήματο. Γιατί πιστεύω πω πολλέ χώρε δεν θα τα καταφέρουν. Μέσω της, ε, των διαρροών ε, του offshore και όλων αυτών των ε, ανακοινωθέντων στον τύπο, η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγής έχει μια νέα ευκαιρία μπροστά τη, γιατί τώρα ξέρουμε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένου φορο ε, διαφύγοντες και αυτό μπορεί να το λειτουργήσει ως ε, κίνητρο να λειτουργήσουν ηθικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπως γίνεται σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Έχω μεγάλο σεβασμό για τη νέα μέθοδο καθονομασίας συγκεκριμένων παρανομιών γιατί αυτό βοηθά, που γίνεται στον τύπο, γιατί αυτό σημαίνει πως θα βοηθήσει στο να επανέλθουν τα χρήματα στις χώρες. Τώρα για το θέμα της νομιμότητας, η συλλογή των φόρων <coughs> μπορεί να βοηθήσει, γιατί όπω σα είπα ο κόσμος του ή άλλω τα συγχαίει όλα αυτά. Πάντω τα χρήματα που συλλέγονται δεν είναι προ όφελο τη συζήτηση κατά του ξεπλήματο του βρώμικου χρήματο και της καταπολέμησης αυτής της ε, κατάστασης. Οι καταδίκες και τα κατησχεμένα χρήματα θα πείσουν τον κόσμο να μετρήσουν ε, βέβαια την επιτυχία αυτών των μέτρων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω σε σχέση με τον κίνδυνο του να υπερβάλλουμε τα νούμερα. Η Γερμανία, ας πούμε, επικρίθηκε γιατί οι σχετικές εκθέσεις δεν ήταν, λέει, αρκετά ψηλές. Εδώ έχουμε έξι, τρεις εκθέσεις και δείχνουμε πως κάθε χώρα θα μπορούσε εύκολα να κάνει δέκα φορές περισσότερες εκθέσεις εκθέσει, φουσκώνοντα τα, τα νούμερα. Νόμιμα και όχι παράνομα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αν έλεγε ο κύριο Δεβάλλοντα τη τράπεζα, μην αναφέρετε μια φορά την ημέρα, αλλά κάθε φορά που γίνεται μια συναλλαγή θα μπορούσε να προσθέσει 3 ή 5 ευρώ, ε, μηδενικά στις γεννημαρικές εκθέσεις. Οπότε σε ορισμένε χώρε ε, η, η, η, η, αναφορά γίνεται σε ομάδες, σε σύνολα, εξαρτάται από την κάθε χώρα. Ε, και δεν θέλουμε υπερβολικά νούμερα για τη Γερμανία, ας πούμε. Η Γερμανία έχει ακολουθήσει κάθε σύσταση, τότε μπορεί να παραπονεθεί ότι αυξήθηκε το ξέβλημα βρώμικου χρήματος αντί να μειωθεί. Τα νούμερα λοιπόν δεν πρέπει να τα δίνουμε μεγάλη σημασία γιατί οι χώρες είναι διαφορετικές. Εγώ ε, πιστεύω με το γερμανικό σύστημα ακόμα και αν τα νούμερα είναι χαμηλά, ενώ με άλλες χώρες δεν θα τις εμπιστευόμουν ό,τι και να κάνουν. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις μαύρες λίστες, αν και οι μαύρες λίστες είναι επιτυχείς, είναι υποπίεση από τις μεγάλες χώρες, δεν αναγράφουν κάθε φορά, δεν τις εμπιστευόμαστε βέβαια απόλυτα γιατί είναι προκατηλημένες. Ένα σημείο είναι ότι ας πούμε η ΕΠΑ ποτέ ούτε καν συζητήθηκε να μπει σε κάποια λίστα μαύρη. Περισσότερο θα πρέπει να εστιάζουμε στις καλύτερες πρακτικές, στις άσπρες λίστες. Το ξέβλημα βρώμικου χρήματο χρειάζεται πραγματική συμμόρφωση. Δεν χρειάζεται να γίνονται τέτοια παιχνίδια νούμερων Πρέπει να πείσουμε τις χώρες, τα Υπουργεία, τα, τους εισαγγελείς, τα δικαστήρια κτλ. ότι είναι ένα σημαντικό θέμα κατά πολέμηση αυτού του εγκλήματος. Επίσης, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, να καταστήσουμε σαφές πως η ισχύ της Ευρώπη δεν είναι το να κάνουμε unisex προσεγγίσεις όπως κάνουν οι Αμερικάνοι. Ε, η Ευρώπη πάντα είναι διαφορετική. Έχουμε ιστορία διαφορετικών θεσμικών και νομικών συστημάτων Έχουμε τον Απολέοντιο κώδικα στην Γαλλία, το Ρωμαϊκό δίκαιο και όλα αυτά δεν ταιριάζουν απόλυτα για να έχουμε το ίδιο στάνταρ. Έχουμε λοιπόν να μελετήσουμε τεσσάρων ειδών Ευρώπες. Η πρώτη είναι αυτοί που ε, έχουν μεγάλες δυσκολίες να εφαρμόσουν συστήματα κατά του ξεπλήματος γιατί το νομικό του σύστημα δεν ταιριάζει, δεν, δεν καλύπτει διπλά, διπλή τιμωρία. Ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες και στην ε, Βόρεια Γερμανία τα νομικά συστήματα έχουν δυσκολίες να σωματώσουν αυτές τα προδιαγραφές. Έχουμε κάποιες χώρες όπου ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν είναι η πρώτη τους προτεραιότητα το ξέπλυμα χρήματος. Πολλές από τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτά τα στάνταρ. Και όταν αντιγράφουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν σημαίνει πως κάτι θα κάνουν κιόλα με αυτή την οδηγία. Έχουμε την Ολλανδία, την Κύπρο και την Λουξεμβούργο που είναι άλλη ομάδα που έχουμε μικρές χώρες που κατακλείζονται από πολύ συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένες καταστάσεις. Ε, όπως είπαμε δεν χρειαζόμαστε ομοιομορφία εδώ <laughs> και σίγουρα δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερα νούμερα ε, και φούσκωμα των αριθμών. Να δούμε κάθε χώρα σε τι είναι καλή πρέπει. Ας πούμε στην Εστονία δεν μπορεί κανείς να πληρώσει μετρητά. Ακόμα και ο ταξιτζής ε, παίρνει μόνο κάρτα. Η Εστονία είναι σχεδόν χωρίς μετρητά. Εάν δεν κυκλοφορούν μετρητά λοιπόν θα αποφύγουμε ένα μεγάλο αριθμό ξεπλήματος, μεγάλο όγκο μάλλον ξεπλήματος μέσω μετρητών. Μπορούμε λοιπόν να μάθουμε και να αναπτύξουμε κάτι που να είναι ένα ευρωπαϊκό στυλ κατά της, ε, του ξεπλήματος και όχι αμερικανικό σύστημα όπου η τιμωρία είναι το πάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ανοίγει η συζήτηση. Δίνω το λόγο στον κύριο Γιακολίνο, τον εισηγητή. E Ακούσαμε και τις τρεις ε, παρεμβάσεις που ήταν άκρος ενδιαφέρουσες και μπορούμε έτσι να λάβουμε υπόψη και τις δικές μας τροπολογίες. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή πρέπει να καταρτήσει μία πρόταση οδηγίας για την ανακύκλωση βρώμικου χρήματος. Εμείς προβλέπουμε στο έγγραφό μας και την ε, αντιμετώπιση της αυτοανακύκλωσης. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να προβλέψουμε και την φόρο αποφυγή και την φόρο ε, διαφυγή και να θεωρούνται εγκληματικές πράξεις, αξιόπινες ε, πράξεις. Ως προς τους ε, φορολογικούς παραδείσους, φαίνεται ότι έχουν κατώτερο αριθμό από τον αρχικά προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν είναι 60. Θα ενημερωθούμε και θα επικαιροποιήσουμε τους καταλόγους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε ένα διπλό νομοθέτημα, το TUPAC, το οποίο θα αποτελέσει βάση και της Τραπεζικής Ένωσης. Τι σκέφτονται οι τρεις εισηγητές. Και ο δημοσιογράφος, τον οποίο ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάγκη άρσης του τραπεζικού απορρίτου εμείς ε, το προβλέπουμε στην πρότασή μας και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι απόλυτα αναγκαίο έτσι ώστε να αρθεί για να ξέρουμε από πού προέρχονται πάντα τα χρήματα, οι εισρωές. Και αυτό αφορά και ορισμένα μεγάλα κράτη-μέλη, όχι μόνο τα μικρά. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Ο κύριος Νιούτον Ντάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις εξαιρετικές ε, παρουσιάσεις. Ε, ευχαριστώ. Στον κύριο Ντεβάου ήταν ένα ερώτημα. Από, αυτά τα, από αυτό το μεγάλο αριθμό εκθέσεων που μας αναφέρατε, μπορεί να είναι και χίλιες φορές περισσότερες ή και λιγότερες, αλλά από αυτές τις εκθέσεις, εν πάση περιπτώσει, πόσες οδηγούν σε δίωξη τελικά και σε τιμωρία γιατί κάθε κράτος μέλος μπορεί να, τα, να συλλέξει τέτοιες εκθέσεις, αλλά υπάρχει κάποια συνέχεια. Δεύτερον, η δική σας σύσταση στη δική μας την Επιτροπή ποια είναι. Τι πρέπει να πούμε στην Κομισιόν να προτείνει ώστε να αλλάξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και σας ευχαριστώ. Τώρα, για τον, Κροατό, για τον ε, δημοσιογράφο. Η Κροατία ακόμη δεν έχει ενταχθεί επισήμω, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε κροατικά, αλλά θα γίνει γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα η ε, παρουσίασή σας. Εσείς κινδυνεύσατε, σας έχουν απειλήσει όταν κάνατε την έρευνά σας, γιατί ήταν επικίνδυνα τα νερά που κολυμπήσατε. Και επίσης και εσείς ε, το ίδιο ερώτημα, τι θα μας προτείνατε στην Επιτροπή μας να κάνουμε και για την ε, κυρία, την καθηγήτρια Ούγκερ. Πολύ χρήσιμε οι πληροφορίε σα. Ελπίζω ότι θα μα στείλετε και τα αποτελέσματα για να τα μελετήσουμε καλύτερα. Δύο σύντομα ερωτήματα. Ένα. Είπατε τέσσερι χώρε μονάχα δεν είναι μέλη της FATF. Ποιε είναι αυτές οι τέσσερι. και οι δικέ σας συστάσει, οι προτάσει σα προ την Επιτροπή μα ποιε είναι. Øh, Ο ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις παρεμβαίνοντες. Σε πολύ ε, ενημερωτικές οι παρουσιάσεις σας. Ελπίζω ότι θα λάβουμε και τα αντίτυπα των ε, παρουσιάσεών σας για να τα μελετήσουμε. Κάτι για την ε, Δόκτωρ Ούγκερ. Κάνατε κάποιες αναφορές σε κάποιες λευκές λίστες θεωρώ ότι είναι καλή πρόταση αυτή και νομίζω ότι όντως και με τις μαύρες λίστες υπήρξαν προβλήματα γιατί είναι πολιτικώς δυνατό να επηρεαστούν αλλά νομίζω ότι ε, πληρούν και κάποιες προποθέσεις αυτές οι λίστες. Ε, δηλαδή, με βάση αυτές τις λίστες κάτι έγινε, παρόλο που βεβαίως οι λευκές λίστες είναι πολύ καλύτερες. Αλλά και πρέπει να δεχτούμε ότι κάπως βοήθησαν και οι μαύρες λίστες. Μετά, ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τις ε, βέλτιστες πρακτικές. Μερικές φορές έχουμε δύο εναλλακτικέ. Καταρχάς έχουμε το νόμο ή το δικαστικό σύστημα και από την άλλη έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, καμιά φορά είναι... Είναι έτσι λίγο ε, ε, χαλαρό ας πούμε το σύστημα αυτό με τις βέλτιστες πρακτικές. Ίσως να θεωρείτε ότι δεν είναι πολύ αυστηρό ή πολύ στέρεο. Εσείς πώς το βλέπετε. Και μετά, ε, για τα όσα είπε ο, κύριος από την ε, Κροατία. Είναι πολύ καλή, πολύ ωραία όλα αυτά που μας ε, παρουσιάσατε, αλλά παρόλα αυτά σκέφτομαι μήπως λείπει κάτι από την όλη ιστορία, γιατί όλα αυτά τα χρήματα, όλες αυτές οι τράπεζες που εδώ και χρόνια χρησιμοποιούνται από το 1995 μέχρι το 2007, και είπατε ότι η κυβέρνηση ήξερε και μάλιστα συμμετείχε. Αλλά υπήρξαν διάφορες κυβερνήσεις σε, σε αυτό το χρονικό διάστημα του 1995 μέχρι το 2007. Υπήρξε αλλαγή στην κυβέρνηση, υπήρξαν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, λαϊκές κυβερνήσεις. Ε, και εδώ μας είπατε ότι ουσιαστικά είτε άλλαζε η κυβέρνηση είτε δεν άλλαζε, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Αν ισχύει αυτό, τότε δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα. Σημαίνει ότι δημιουργήθηκε ένα σύστημα το οποίο ήταν τελείως ανεξάρτητο από, το, από αυτούς που το, που το εξέλεξαν και από αυτούς που το ήλεγχαν. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται, τι κάνει κανείς με αυτά τα χρήματα. Και επίσης κάτι άλλο εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ακόμη τέτοια χρήματα από τέτοιες δραστηριότητε στην Κροατία σήμερα και επίσης η Κροατία με, ε, έχοντας και το, την προοπτική ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανεχθεί τέτοιες ε, υποθέσεις. Αυτό είναι τεράστιο ερώτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι βέβαια και θέμα πολιτικού πλαισίου και είναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις σας και σας ευχαριστώ πολύ για το όσα μας είπατε. Ο κύριος Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντεβάλ. Να μας πει πώς ε, μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ε, ανακύκλωση. Δηλαδή, γιατί αριθμητικά ε, στοιχεία μιλάμε ως προς τη ροή κεφαλαίου, ιδιαίτερα από την παράνομη εμπορία και ιδιαίτερα ως προς τα ναρκωτικά. Και Πώς μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε τα στοιχεία. Πολλοί εμπειρογνώμονες μας λένε ότι δεν ε, μπορούν να ανακυκλωθούν τεράστια κεφάλαια χωρίς να, υπάρχουν, ε, χωρίς να υπάρχει το στήριγμα και υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος. Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε εσείς Εδώ μιλάμε για Ρώσους, Τούρκους και ούτω καθεξής. Ε, γίνεται λόγος και για την Ιταλική μαφία. Στη Γερμανία υπάρχει Ιταλική μαφία. Ε, έχει ε, με βάση ε, τη, τα διάφορα δεδομένα, πληροφορίες και ούτω καθεξής. Γιατί από το Ιταλικό παρατηρητήριο και από τα δικά μας ε, ε, και από τις δικές μας ε, αστυνομικές και δικαστικές αρχές προκύπτουν πολλά στοιχεία για τη διείσδυση της μαφίας. Θυμάμαι μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που μου ελέγχθη. Ένας μεγάλος ιστορικός μου είπε ότι στα γερμανικά, ε, από τα γερμανικά αρχεία, ακόμα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η καμόρα ε, μπορούσε να επιδοθεί σε εμπόριο. Υπήρχε ένα ευρύ δίκτυο. Νομίζουμε λοιπόν ε, μιλάμε για μια ελεύθερη οικονομία και ε, δεν μιλάμε για, ε, βεβαίως εδώ, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά για τους ελέγχους, διότι μετά από την μεγάλη κοινή σφαγή δεν είχαμε εμπεριστατωμένες μελέτες για αυτό το μεγάλο ε, Ιταλικό καρκίνωμα, δηλαδή το καρκίνωμα της Ιταλικής ε, μαφίας στη Γερμανία. Ως προς την ε, Κροατία θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την έρευνά σας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ανοιχνεύεται αυτή η δραστηριότητα πάντα και θα πρέπει να γίνονται οι σωστοί συσχετισμοί και να προωθείται ο διάλογος με τις ερευνητικές αρχές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω έρευνας, γιατί μιλήσατε για ροή κεφαλαίων, για την ανόρθωση της οικονομίας, παγκόσμια τράπεζα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές γίνονται προς ε, υποψήφιες χώρες και ποια είναι η έκβαση. Πώς ε, έχουν σήμερα οι έλεγχοι έτσι ώστε να αποφευχθούν ε, τέτοιοι κίνδυνοι. Έχει μεγάλη σημασία. θα πρέπει να δούμε τι ενδείξεις έχουμε και τι ενδείξεις έχει η Όλαφ. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο. Σας υπενθυμίζω στα πλαίσια της ε, συζήτησης ε, πρώτα έχουν το λόγο οι συντονιστές, ε, οι συζητητές και μετά οι βουλευτές. Βάιλερ. Το καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε αλλά εγώ εκπροσωπώ τον συνάδελφο από τους σοσιαλιστές. Ε, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ε, είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, το ε, πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με, τον, ε, τα όσα είπε ο δημοσιογράφος από την Κροατία. Στην, με την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς πήγαμε στην Κροατία για να δούμε πώς λειτουργεί η νομοθεσία σήμερα, πώς λειτουργούν τα τελωνία, τι γίνεται με τις δημόσιες συμβάσεις και είχαμε την εντύπωση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά πράγματα στην Κροατία. Γι' αυτό το ερώτημα μου προς εσάς είναι το εξής. Έχετε την ε, ε, εντύπωση ότι έχουν όντως διακπεριωθεί κάποια πράγματα, ότι εκεί που οι ένοχοι ε, τιμωρήθηκαν τα χρήματα ανακτήθηκαν, υποθέτω ότι το παρακολουθείτε, οπότε θα ήταν και για μας πολύ ενδιαφέρον. Παρόλο που δεν αλλάζει τίποτα για την ένταξη της Κροατίας, η Κροατία θα έρθει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξέρουμε, να μας πείτε αν όντω έχει αλλάξει κάτι και η κατάσταση τώρα πώς έχει. Στο παρελθόν ακούσαμε, και εσείς θα το ξέρετε, ότι και η Γερμανία ήταν, είχε εμπλακεί με μια τοπική ε, τράπεζα σε ένα κρατήδιο σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο με την Χύπο. Ε, οπότε ερωτώ, ε, έχετε δει βελτίωση στην Κροατία. Δεύτερο ερώτημα στους άλλους δύο ομιλητές, κυρίως στην Δόκτωρ Ούγκερ. Έχω, άκουσα κάποια αντίφαση. Από τη μία είπατε ότι είναι πολύ χρήσιμο το να καταδεικνύει κανείς ποιος φταίει ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιους τομείς. Το χρησιμοποιούμε. Ε, βεβαίως καταδεικνύουμε και, τους, και όσους τα πάνε καλά, όχι μόνο τους κακούς, εισαγωγικά. Και όσα έχει τέτοιες λίστες που, λένε ότι, που λέει σε αυτές τις, αυτές χώρες πάει καλά η αντιμετώπιση διαφθοράς και σε αυτές όχι. Απ' την άλλη είπατε ότι οι μαύρες λίστες είναι κακές, είναι κακή επιλογή. Οπότε πού είναι η διαφορά, θα θέλαμε, να μου το διευκρινίσετε λίγο. Και ένα δεύτερο. Ε, και εγώ όπως και εσείς πιστεύω ότι η δημοσιομική κρίση ήταν πραγματικά μια, ε, ε, ένας κινητήριος μοχλός που ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή για όλες τις χώρες και στο Λίχτενσταϊν και στην Αμερική και σε άλλες οάσεις Νομίζω όμως ότι το καλό είναι ότι ε, ασχολείται πια η κοινή γνώμη με αυτό. Δεν ασχολούνται μόνο οι διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί, αλλά και στους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα από αυτήν και έξω από αυτήν. Ασχολούνται, υπάρχουν ε, διαδηλώσεις, ε, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει πια αποδεκτό αυτό, η, το ξέπλυμα μαύρου χρήματο η αποφυγή, η απάτη, όπως ε, παλιότερα. Τώρα πια αναγνωρίζει κανείς ότι λείπουν χρήματα από το κράτος. και ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι να μειώνονται τα κοινωνικά επιδόματα για να ξαναγεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Οπότε για μένα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω την απόψή σα. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τον Γερμανό εκπρόσωπο. Όπω και εσεί και η κυρία Όγκερ, και εγώ θεωρώ ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι το παν ούτε ε, το να έχουμε ποσοτικά στατιστικά μας ε, βοηθάει. Θέλουμε ποιοτικά στατιστικά προφανώς, αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν έχετε κι εσείς την εντύπωση ότι τελευταίως στη Γερμανία, ε, λόγω και της συζήτησης που διεξάγεται, ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα στην Γερμανία, ότι δηλαδή έχουμε πολύ κατεγραμματισμένες δομές σε κρατήδια, που πρέπει να δαπανίσουν το κόστος της ε, έρευνας και στο τέλος δεν μπορούν να κρατήσουν ε, τα χρήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχέσουν ότι πρέπει να τα, να τα αποστείλουν ας πούμε στις κεντρικές αρχές. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα αρμοδιοτήτων βεβαίως. Ε, πολλές φορές έχουμε πει ότι υπάρχουν πολλές δομές και υπάρχουν επικαλύψεις και καμιά φορά είναι και ανεπαρκείς αυτές οι δομές. Και κάτι τελευταίο. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δυνάμεις της και με την ε, με τις πολιτικές δυνατότητες που έχει μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε αυτό το θέμα της διαφθοράς, του ξεπλήματος. και της φοροαπάτης. Είσαστε και εσείς της άποψης ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εισαγγελία έτσι όπως την σχεδιάζουμε. Βεβαίως έχοντας υπόψη πάντα ότι Κάποιες χώρες έχουν διαφορετικές ε, νομικές παραδόσεις, αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε ότι ε, τα εγκλήματα είναι διασυνοριακά. Δεν περιορίζονται μόνο σε περιφέρειες ή σε κράτη. Οπότε θα ήταν λογικό ίσως και σκόπιμο να προχωρήσουμε κι εμείς με ένα πιο διασυνοριακό μοντέλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βάλερ. Η γραμματεία μου έλεγε πως δεν έχει φτάσει κάποια ανακοίνωση από την κύριε Φαγιόν. Αν θέλετε λοιπόν στείλτε μας ώστε να το έχουμε κι εμείς. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους εισηγητές μας για να δώσουν τις απαντήσεις τους. Θα συνεχίσουμε με τη σειρά με την οποία ξεκινήσαμε, ο κύριος Ντέλβαλτ, μετά ο κύριος Μάρια και μετά η, κυρία, η καθηγήτρια Ούγκερ. Ο κύριος Ντεβάλτ πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Το πρώτο ερώτημα που μου τέθηκε ήταν ποιες είναι οι βελτιώσεις που βλέπει κανείς, κυρίως για το τραπεζικό απόρριτο. Πώς έχουμε αλλάξει τα πράγματα, αν έχουμε βελτιώσει τα πράγματα. Αυτό άπτεται ενός πολύ μεγάλου προβλήματος. Γιατί ξεπερνά το τραπεζικό απόρριτο. Πάντα όταν χρειαζόμαστε πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες δεν είναι είτε αξιόπιστες είτε δεν έρχονται έγκαιρα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί και για την αντιμετώπιση της, ε, ε, του ξεπλήματος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι προφανώς ε, ε, διακρατικό και αρκετά ρευστό, αρκετά δυναμικό. Αν εγώ, ε, αν εμένα μου είχαν κάνει ένα έμβασμα πολλών εκατομμυρίων στο λογαριασμό μου, την επόμενη ώρα θα μπορούσα να χωρίσω το ποσό αυτό σε μικρότερα, να το στείλω παντού στον κόσμο και να μην το βρει κανείς. Υπάρχουν ε, ε, πολλά φόρα, πολλά βήματα που ασχολούνται με ε, οικονομικές υπηρεσίες. Μπορεί κανείς λοιπόν να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες ακόμα και για σήμερα ας πούμε να αγοράσει μια επιχείρηση να, και όσο πιο πολύ επενδύει εγώ, α πούμε, έχω μια επιχείρηση και σήμερα το απόγευμα, μόλι πάω σπίτι μου, θα μπορούσα να αγοράσω 12 επιχειρήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Χωρί καν να χρειαστεί να ε, επενδύσω πάρα πολύ. Χρειάζομαι κάποια ευρώ και χωρί πρόβλημα, χωρί πρόβλημα όμω, μπορώ να αγοράσω τέτοιε επιχειρήσει. Είναι δηλαδή ένα all-included ε, πακέτο. Μπορείτε να το δείτε κιόλα ε, σε ποιε δικαιοδοσίε μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι λοιπόν αρκετά εύκολο σήμερα ειδικά να γίνει αυτό. Και επίσης θα μπορούσα να, σήμερα το βράδυ να είμαι και διευθυντής τράπεζας. Εντάξει, θα μπορούσα, θα χρειαζόταν βεβαίω να επενδύσω λίγο περισσότερο από καμιά εκατοστή ευρώ, αλλά άμα α πούμε με ένα πενταψήφιο νούμερο, εύκολα θα μπορούσα να γίνω το βράδυ διευθυντή τράπεζα. Αυτό είναι βασικά το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ότι το έγκλημα κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Για να μπορέσουμε λοιπόν εμεί οι διεκτικέ αρχές να κινηθούμε λίγο πιο εύκολα, χρειαζόμαστε και σε σχέση με αυτό που κάνει και η FATF, ε, χρειαζόμαστε λοιπόν τραπεζικά δεδομένα. Στη Γερμανία έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία, γιατί έχουμε ένα κεντρικό μητρό τραπεζών. Και σε σχέση με αυτό που είπε και η δόκτωρ Ούγκερ, αυτή είναι βέλτιστη πρακτική. Δεν θα βρείτε κανέναν από τις διοικητικές αρχές που θα σας πει ότι δεν είναι χρήσιμο αυτό. Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ εντάξει, να μην πω σε πολλέ λεπτομέρειε, αλλά υπάρχουν και άλλα μητρώα ή θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα α, μητρώα τα οποία θα διευκόλυναν πάρα πολύ τη ζωή των διοκτικών αρχών πραγματικά πάντα διαπιστώνω με μεγάλη έκπληξη ότι δεν χρειάζεται καν να πάμε εκτός Ευρώπης. Και εντός της Ευρώπης υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα. Ας πούμε, αν δούμε ότι στην Ισπανία σε μια ε, μεγάλη δράση που έγινε πριν από λίγα χρόνια το οργανωμένο έγκλημα, ε, κατασχέθηκαν μάλλον από οργανωμένους εγκληματίες ε, πάρα πολλά ε, ε, περιουσιακά στοιχεία, πάρα πολλά κτίρια, θα μπορούσε να υπάρχει ας πούμε ένα μητρό τέτοιων κτίριων που μπορούν να ανακτηθούν. Γιατί να μην υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει ένα μητρό κεντρικό για τις ασφάλειες. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να μας διευκολύνουν τη ζωή. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές περίπλοκες δομές κτλ. Τα πράγματα είναι απλά. Αλλά δυστυχώ το απλό είναι το δύσκολο να εφαρμοστεί συνήθω. Δεύτερον, αναγνώριση, ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση είναι το σημείο κλειδί. Κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με συναλλαγές. Γιατί αν ε, δεν ξεκινάει αυτό με έναν ε, πολύ τυπικό τρόπο από το κράτος, ούτε εμείς οι ιδιωτικές αρχές μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί. Γι' αυτό είναι κεντρική ουσιώδου σημασία το θέμα αυτό και βεβαίω έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση που έγινε ε, παλαιότερα και θα ξαναγίνει κυρίω για, τα για τα ηλεκτρονικά εργαλεία πληρωμή. Όπου εκεί υπάρχουν όλο και, περισσότερο, όλο και πιο καινούργια μέσα. Αν δείτε λοιπόν ότι μπορούμε, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ε, δυνατότητες θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία ταυτοποίησης. Και υπάρχουν ε, πάρα πολλές εξαρτίες marketing που μπορούν να κάνουν τέτοιες δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει κανείς ε, πληροφορίες, ένα, τηλεφωνο, ένα νούμερο τηλεφώνου ή ένα email Αλλά δεν μπορεί κανείς να στέλνει τέτοια α, στοιχεία προσωπικά του δεδομένα σε μη αξιόπιστες πηγές. Και κάτι τελευταίο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η FATF κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και η ε, Dr. Unger το είπε, έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα σε αυτόν τον κόσμο της αξιολόγησης, Βεβαίω, οι, οι μονάδε για την αντιμετώπιση του ξεπλήματο δεν υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάνει κάποια βήματα Και εν τω μεταξύ δεν θα δείτε κανένα κράτος στον κόσμο που να έχει ολοκληρώσει το σύστημά του. Το πρόβλημα που έχουμε είναι εφαρμογής, πρόβλημα εφαρμογής και γι' αυτό προσπαθούμε να το, να το δούμε πιο προσεκτικά. Και θα κλείσω εδώ κάνοντας κάποιες προτάσεις. Μίλησα πριν για ταυτοποίηση. Αυτή είναι μία πτυχή. Αλλά ποιο είναι ο δικαιούχο. Αυτό είναι η άλλη πτυχή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ταυτοποίηση και μετά να μπορούμε να παρακολουθήσουμε ότι ε, θα δημοσιοποιείται ας πούμε και το όνομα του δικαιούχου. ο οποίο θα μπορεί να συλληφθεί, θα μπορούν να γίνουν ε, ανακρίσει, θα μπορεί να εμπλακούν οι ιδιοκτικέ αρχέ όλα αυτά θα πρέπει να μπορούν να γίνουν, γιατί το πρόβλημα υπάρχει. Μετά, κάποια άλλα ερωτήματα που μου τέθηκαν για την επιτυχία των ε, ε, εκθέσεων που λαμβάνουμε. Και ευχαριστώ βεβαίω και την ε, κυρία Ούγκερ. Όντω, η ποιότητα δεν, η ποσότητα δεν σημαίνει και ποιότητα. Ναι, είναι ε, καλές οι εκθέσεις ως προς την ποσότητά τους, να μπορεί κανείς να δει μέσα από πολλές ε, συναλλαγές μεμονωμένες ας πούμε και να τις αποστέλνει ως συγκεκριμένες δηλώσεις αλλά υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Για, κάθε, για κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε εμείς τη θεωρούμε ως μεμονωμένη περίπτωση όσο μικρή και, ή μεγάλη κι αν είναι. Και αυτές οι ε, δομές που έχουμε οδηγούν τελικά σε έρευνες. Δεν έχω τώρα τα στατιστικά υπόψη μου, αλλά μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας και στην ετήσια έκθεση, μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά στοιχεία. Ήδη από το 2002 5 ή 6 ή 7% σίγουρα κάτω από 10% των περιπτώσεων κάνουμε, ε, ε, έτσι, παραγράφονται ας πούμε κάποιες, ε, κάποιες υποθέσεις. Οι υπόλοιπε θεωρούνται με περιπτώσεις και οδηγούν συνήθως σε δίωξη. Μετά, το επόμενο ερώτημα. Για τις προτάσεις βελτίωσης. Είπα κάποια πράγματα. Να σας αναφέρω και το έγγραφο που υπήρξε από την FIU προς την Κομισιόν και τα 27 FIUs το συμφώνησαν το κείμενο αυτό και είπαμε ότι στο μέλλον θα ήταν καλό να υπάρχει μια σχετική οδηγία από την Κομισιόν. Μετά, μου ετέθηκε το ερώτημα τι γίνεται με τον όγκο του ξεπλήματος Ο όγκο με τον, οποίο, έχουμε, να κάνουμε στη Γερμανία, για το ξέπλυμα συγκεκριμένα, δεν, δεν μπορεί να υπολογιστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπολογισμό δηλαδή, εκτίμηση ε, του, του, όγκου το, που βρίσκεται, του όγκου του που βρίσκεται εντός Γερμανίας και εκτός βεβαίως. δεν είναι δυνατόν να υπολογίσουμε ε, ούτε καν εντό Γερμανία πόσο είναι ο όγκο των χρημάτων, γιατί ε, μπορεί κάτι να γίνει ε, μέσω Γερμανία ή μπορεί να υπάρξουν χρήματα που, μαύρα χρήματα από, από άλλη χώρα εκτό Γερμανία που να επενδυθούν με κάποιο τρόπο στη Γερμανία. Οπότε αυτό είναι δύσκολο να το εκτιμήσουμε. και όποιος ε, θέλει να δράσει θα πρέπει να παραδεχτεί ότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό, ότι τελικά δεν είναι δυνατό ε, να υπολογιστεί όγκος αυτός. Η Ιταλική μαφία στη Γερμανία. Εδώ μιλούμε για ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρείται εδώ και χρόνια. Στην αρχή της παρουσίασής μου έκανα μια έτσι, εμπαρόδο παρατήρηση για το ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσα να βάλω και στοίχημα ότι στις επόμενες εβδομάδες το ξαναδούμε και στα ΜΜΕ για το πόσα περιουσιακά στοιχεία ε, της Ιταλικής μαφίας ε, περνάνε από την Γερμανία ή επενδύονται στη Γερμανία. Αυτό που μπορώ να σας πω, και ξέρω ακριβώς τι λέω, γιατί εγώ είμαι παρόν σε τέτοιες συζητήσεις, με, την Ιταλ... με τους Ιταλούς συναδέλφους ε, συναντιόμαστε συχνά, συζητάμε εντατικά, έχουμε πολύ επαγγελματική ανταλλαγή απόψεων και κάθε φορά λέμε ότι σας παρακαλούμε όταν έχετε τέτοια στοιχεία και τα είναι, είναι συγκεκριμένα και επίκαιρα, στείλτε τα μας και κάθε, κάθε, τέτοια, κάθε δήλωση ή πληροφορία που μας δίνεται την παρακολουθούμε με, μεγάλο επαγγελματισμό. Τώρα, τα παραδείγματα που είπατε και το πιο σημαντικό ήταν τα στατόπεδα συγκέντρωσης. Το ξέρουμε βεβαίως και από τις τρέχουσες καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο να ελέγξουμε τέτοιες περιπτώσεις. περιπτώσεις. Ακόμα και σε σοφρονιστήρια είναι δύσκολο. Ακόμα παντού στον κόσμο είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να, αντιμετωπίσουμε το εμπόριο ναρκωτικών είναι πάρα πολύ περίπλοκο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώ σε μια ανοιχτή κοινωνία που όλοι θέλουμε και για όλοι αυτήν προσπαθούμε, ε, είναι απολύτω. αδύνατο. Τώρα το πόσο θα ανεχθούμε το ξέπλυμα χρήματος κτλ ή πόσο μπορούμε να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες δράσης στις, α, αρχές, αυτό μπορούμε να το δούμε. Αλλά από τη μία θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, από την άλλη θέλουμε όμως να έχουμε και ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και κεφαλαίων και αγαθών. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ε, είναι εκνευριστικό το ότι δεν προχωρούν, γιατί εκεί όντως θα θέλαμε πιο συγκεκριμένα, πιο ισχυρά εργαλεία. Αλλά δεν, δεν πιστεύω ότι οι περιορισμοί, γιατί όλοι οι πολίτες είμαστε, και μπορεί να, κάποια στιγμή να είμαστε εμείς το αντικείμενο μιας έρευνας. Ε, θα πρέπει να περιορίσουμε τα ε, δικαιώματά μας για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν τα δεδομένα αυτά ε, τηρούντο, αποθηκεύονταν για πολύ περισσότερο όταν κάνουμε τέτοιες ε, έρευνες, να μπορούμε δηλαδή να ε, χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους δεδομένα. Και ξαναέρχομαι σε αυτό που είχα πει στην αρχή. Όταν κάνουμε έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, Συνήθω αυτό γίνεται με καθυστέρηση, χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή παίρνουμε τι πληροφορίε αφού έχει υπάρξει, έχουν υπάρξει πολλέ πληροφορίε, έχουν υπάρξει ενδείξει και ο κύριο δίπλα μου δημοσιογράφο δεν μπορεί τώρα που παίρνει την πληροφορία τώρα να ε, φτάσει στην διοκτική αρχή. Ε, πολλέ φορέ είναι έτσι μια αίσθηση που έχει κανείς, μετά ακούει κάποια πράγματα, μετά λαμβάνει πληροφορίε πληροφορίες και πολύ αργότερα ξεκινάει η έρευνα. Οπότε, αυτά τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, όταν δεν μπορούμε να τα έχουμε ή όταν δεν, μπορούμε, ε, δεν είναι πια αποθηκευμένα και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί κάποια κράτη-μέλη ε, δεν αποθηκεύουν αρκετά, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τέτοια δεδομένα και τα δεδομένα εξαφανίζονται, προφανώς για μας είναι αδύνατο, αδύνατο να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε ε, τις έρευνές μας. Οπότε πραγματικά θα ήθελα να υπάρξει μια εναρμόνιση ως προς αυτό στην Ευρώπη για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα με τέτοια, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια δεδομένα για περισσότερο χρόνο. Ε, κατάδειξη, ναι, των κακών σε εισαγωγικά, ε, βέλτιστες πρακτικές από την άλλη. Οι βέλτιστες πρακτικές προφανώς είναι πολύ σημαντικές. Πιστεύω ότι συνολικά ε, μπορούν να λειτουργήσουν και ως κίνητρο για να δούμε τι είναι καλό και τι λειτουργεί σε ό,τι αφορά την, το ξέβλεμα μαύρου χρήματος, αλλά ε, βεβαίως ε, ίσως καλό να θα ήταν να καταγράφουμε και πού ε, υπάρχουν ελλείψεις, πού υπάρχουν προβλήματα. Ας πούμε στην ομάδα Egmont είχαμε προβλήματα με ένα κράτος μέλος, το οποίο λόγω του τραπεζικού του απορρίτου δεν έδινε τα, ε, δεδομένα που χρειαζόντουσαν για μια διεθνή έρευνα. Ε, υπήρξε λοιπόν από την ομάδα Egmont ε, πίεση προς αυτό το κράτος μέλος και τώρα έχουμε φτάσει περίπου στο τέλος της υπόθεσης αυτής έτσι ώστε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και Βεβαίω, καμιά φορά είναι καλό να, να καταδεικνύεται τι εμποδίζει την διαδικασία. Τελευταίο ερώτημα για τις δομές στη Γερμανία το ομοσπονδιακό μας κράτος όντως έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά καλό, έχει αρκετά καλές δομές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα, να τα ενώσουμε όλα σε μία κεντρική ε, μονάδα, γιατί αν γίνει αυτό πάλι θα πρέπει να έχουμε μεμονωμένες ε, υπηρεσίες. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μία υπηρεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν εντός αυτής και κάποιες ε, υπηρεσίες ομάδας, οπότε πάλι θα πρέπει κανείς να συναντάται με διάφορους, διάφορες μονάδες και ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε τώρα. Οπότε σε αυτή την ομοσπονδιακή δομή ε, όπως την είπατε. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ καλές δομές. Έχουμε πολύ καλές ε, μονάδες λοιπόν ε, που συναντώνται, ανταλλάσσουν πληροφορίες, έχουμε διάφορες ε, επιτόπου ε, αστυνομικές υπηρεσίες και τοπικές και ανακρατήδιο. Επίσης έχουμε συνεργασία και με τις ε, φορολογικές αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε βρει κάποιους καλούς δρόμους για να προχωρούμε για να ανταλλάσσουμε πληροφορίε με τι εμπλεκόμενε αρχέ. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Νομίζω αυτά ήταν τα ερωτήματα για μένα. Α, είχατε πει και κάτι άλλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν κοινέ δομές, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινοί δρόμοι ε, δράσης και ακριβώς όταν βλέπουμε κάποια προβλήματα, ίσως να είναι πιο ευέλικτο το σύστημα για να βελτιώσει τις δράσεις του. Θυμάμαι όταν ε, υπήρχε ε, πρώτη φορά, όταν ε, τέθηκε στο τραπέζι πρώτη φορά η ιδέα των κοινών επιχειρησιακών ομάδων. Ε, για να, διευκολυνθούν, να διευκολυνθεί η δουλειά των ε, ε, διοκτικών αρχών διασυνοριακά. Στην αρχή υπήρχαν τεράστιες επιφυλάξεις, μανέα δομή και άλλες απαιτήσει και άλλα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν και άλλα σημεία που πρέπει κανείς να προσέχει. Πώς θα γίνει αυτό. Στην αρχή ήταν όλοι πολύ αρνητικοί απέναντι σε αυτή την ιδέα. Μετά πέρασαν κάποια χρόνια και αυτό το εργαλείο ε, άρχισε να γίνεται λίγο πιο φιλικό προς τους χρήστες, άρχισαν να το χρησιμοποιούν και τελικά είναι καλό να... να δημιουργούνται τέτοιες τυποποιημένες δομές οι οποίες να μπορούν ε, να μας διευκολύνουν την καθημερινή μας δράση έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εντός της Ευρώπης για να αντιμετωπίσουμε ε, το ξέπλυμα χρήματος. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση ήταν το θέμα του τραπεζικού απορρίτου που αναφέρθηκε σε μια από τις ερωτήσεις του Ευρωβουλευτού. Να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι αυτή τη στιγμή είμαι στα δικαστήρια υπόδικος στην Κροατία επειδή αποκάλυψα τραπεζικό απόρριτο. Η υπο Άλπε Άντρια με κατηγορεί ε, και κινδυνεύω με φυλάκιση επειδή αποκάλυψα ένα τέτοιο έγκλημα. Είναι τόσο αλαζόνες. Κοιτάξτε, αυτό το έγγραφο είναι η αποδοχή της Hippo Alpe Andria Group στην Κροατία ότι όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα και τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί για αυτό το σκάνδαλο είναι αληθινά και ακριβή αλλά είναι τραπεζικό απόρριτο. Καλύπτεται από το τραπεζικό απόρριτο και γι' αυτό πρέπει εγώ να τιμωρηθώ ω δημοσιογράφο. Είναι προφανέ ότι κάτι πρέπει να γίνει με το τραπεζικό απόρριτο, ώστε να ρυθμιστεί διαφορετικά. Γιατί διαφορετικά δεν θα μιλά πλέον κανεί για τη διαφθορά στο μέλλον. Δεν θα έχουμε δημοσιογράφους που θα ανακαλύπτουν αυτά, αποκαλύπτουν μάλλον αυτά τα σκάνδαλα διαφθορά γιατί θα φοβούνται την φυλάκιση. Και αυτή αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κροατία. Κανένα δεν ε, στάθηκε μπροστά να πει να προστατευτούν οι δημοσιογράφοι και οι καταγγελτε στην ε, Κροατία όταν μιλάνε για τη διαφθορά, αλλά προστατεύουν την ε, Αλπε Άντρια. Ούτε ένας, ένας, μια δίκη κατά της Χίπο Άλπε Άντρια για πλήσιμο, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή τη διαφθορά ούτε κατά ηθινόντων του ομίλου αυτού. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς εξακολουθούν να διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ σαν να μην τρέχει τίποτα. Μόνο λοιπόν ε, ε, εσείς μπορείτε να ε, νομοθετήσετε διαφορετικά. Κυρίως γιατί η Κροατία θα μπει στην Ένωση μετά από την 1η Ιουλίου και ε, οποιαδήποτε δική σας απόφαση θα είναι υποχρεωτική για την Κροατία. Αυτά λοιπόν για το τραπεζικό απόρριτο. Καλύπτουν, καλύπτει τεράστια διαφθορά και έγκλημα αυτό το ε, ε, τραπεζικό απόρριτο. Ένας ευρωβουλευτής με ρώτησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στην Κροατία <laughs> να αποκαλύψουν τέτοιες υποθέσεις. Φυσικά είναι επικίνδυνο στην Κροατία να πει κανεί την αλήθεια. Εγώ πολύ συχνά λέω ότι η αλήθεια είναι η φθηνότερη στην Κροατία ε, ενώ το ψέμα είναι το ακριβότερο. Άμα λες ψέματα, γράφεις ψέματα, πληρώνεσαι πλουσιοπάροχα στην Κροατία. Ενώ άμα αποκαλύπτει σκάνδαλα όπως για την Χίπο Αλπεάντρια, δεν πληρώνεσαι ή πληρώνεσαι ισχνά. Στην Κροατία δεν έχουμε κανένα είδος προστασίας από τις αρχές. Δεν υπάρχει νόμος για την προστασία για την προστασία των δημοσιογράφων ή των καταγγελτών ή κάποια νομοθεσία που να προστατεύει τους δημοσιογράφους σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ το ζήτησα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ε, πριν από μια, ένα χρόνο να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει τέτοιο είδου νομοθεσία για την προστασία των δημοσιογράφων που μιλούν για την ε, διαφθορά και είπαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και μηχανισμοί για να προστατεύεται ο ερευνητικό δημοσιογραφισμό όταν αποκαλύπτει σκάνδαλα και Τα υποσχέθηκε πριν από ένα χρόνο, τώρα ε, ούτε καν λόγο δεν κάνει γι' αυτό. Ούτε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση κάνει λόγο για όλα αυτά. Κανένα διάλογο δεν έχουμε μαζί του. Γιατί Έτσι φτάνουμε και στο ερώτημα του Ευρωβουλευτή Ζόντεργκάρντ. Κάτι λείπει από την προηγούμενη μου ιστορία και το βασικό είναι ότι είναι η ίδια ομάδα ανθρώπων. Όλοι έχουν ε, φάει από την ίδια πίτα. Σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε τον Πρωθυπουργό, το οποίο ο αδελφός ακριβώς πριν από τις εκλογές έλαβε ύποπτη ε, πίστοση από την ε, τράπεζα LHB ε, που είναι στο λίστα του σκανδάλου. Και μάλιστα πήρε αυτό το εμπίστοση, πήρε αυτό το δάνειο και ο πρόεδρος αυτής ήταν πρώην πρόεδρος της ΧΥΠΟ Γκράμπ στη Ζάγκρεπ. Την, της καπούλαρε από το Ζάγκρεπ και έγινε πρόεδρος της LHB μετά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο τωρινό Υπουργό Δικαιοσύνη συνδεόταν με τα σκάνδαλα της ΧΥΠΟ μέσω της ΛΟΠΑ Press Holding, ενός από τους ομίλους μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Κροατία ήταν μέσα στην, ε, σε, σε σκάνδαλο εξαγοράς ε, από την Europa Press Holding, ενός μεγάλου δηλαδή ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, ο υπουργό που είναι υπεύθυνο για την αστυνομία, ο υπουργό ιστορικών ήταν διευθυντής, ένας από τους διευθυντές, ήταν μέλος δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου του Europa Press Holding, του, του ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώσο αυτός ο όμιλος ήταν μέσα στα σκάνδαλα της Χίπο Αλπε Άντρια. Δηλαδή, Δύο βασικοί υπουργοί που κανονικά θα έπρεπε να ερευνούν τα σκάνδαλα, ο ένας υπουργός δικαιοσύνης, ο άλλος υπουργός εσωτερικών, είναι άμεσα αναμεμειγμένοι στα ίδια σκάνδαλα, οπότε δεν μπορείτε να αναμένετε ότι θα κάνουν οποιοδήποτε είδους έρευνα κατά της ε, το ομίλου αυτού. Επίσης ο Υπουργό Οικονομίας κάποια φάση ασκούσε πίεση υπέρ της ΧΙΠ ε, ο όταν η BLP ε, αγόρασε την τράπεζα αυτή και έπρεπε να διωθεί ε, ε, έγκριση από την Εθνική Τράπεζα της Κροατίας για να αγοραστεί, εξαγοραστεί αυτή η τράπεζα και δεν ήθελε να δώσει αυτή την έγκριση γιατί ήδη υπήρχαν ενδείξεις για ξέπλυμα και οργανωμένο έγκλημα. Υπήρχαν διάφορες εκθέσεις από διάφορες επιθεωρήσεις ε, ε, για το ξένο συνάλλαγμα αλλά ο κύριος Λίνιτς που είναι αυτή τη στιγμή υπουργό Οικονομίας ε, στη Σοσιαλδημοκρατική Κυβέρνηση ήταν ένας από αυτούς που ένας λομπίστας υπέρ του ομίλου Χίπο Αλπεάντρια ώστε να πάρει την έγκριση αυτή από την Εθνική Τράπεζα της Κροατίας. Αφού ήρθε στην θέση του Υπουργού Οικονομίας πριν από ένα χρόνο, διόρισε έναν από τους πιο σημαντικούς του συνεργάτες, έναν άνθρωπο που ήταν ο κύριος υπεύθυνο που συγκάλυψε τα σκάνδαλα ε, της ΧΥΠΟ, ήταν επικεφαλής της ε, οικονομικής επιθεώρησης και τώρα είναι κύριος συνεργάτης του κύριου Λίμιτσης στη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Νομίζω πως αυτό σας τα εξηγεί, κύριε Ζόντεργκάρντα. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία στήριξη, όπως καταλαβαίνετε από αυτή την πολιτική κατάσταση. Δεν έχουμε στήριξη ούτε από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, εγώ συνεργάστηκα μαζί τους και με την ειδική ε, εισαγγελία κατά της διαφθοράς που λέγεται Ούσκο στην Κροατία από το Μάρτιο του 2008 συνεργάστηκα μαζί τους. Ήταν το πιο το σημείο που τους έδωσα τα έγγραφα για την υπόθεση Σενάρκ που έλαβε δωροδοκία από την ε, Όμιλο Χ κατά τη διάρκεια του πολέμου και όπως ίσως γνωρίζετε χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να δραστηριοποιηθεί αυτή η υπόθεση, να ενεργοποιηθεί μάλλον. Είχαν όλα τα έγγραφα στα χέρια τους, απλώς δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα μέχρι ότου να έρθει η κατάλληλη πολιτική στιγμή. Τότε το έκαναν, τα ίδια και τώρα. Τίποτα από τα, κανένα από τα σκάνδαλα του ομίλου Χίπο στην Κροατία δεν διώκεται ποινικά. Ούτε μια υπόθεση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο στην υπόθεση Χίπο στην Κροατία. Και αυτό οφείλεται σίγουρα στον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Μάλιμαϊτς. Αν δεν μπορεί να διώξει ποινικά, ας το πει δημόσια. Ποιος δεν τον ακούει, το Κοινοβούλιο που είναι υπεύθυνο για σένα, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά αυτός πρέπει να το πει δημόσια. Γιατί δεν κάνει τίποτα, γιατί δεν διώκει ποινικά την χήπο για τα σκάνδαλα. Μιλάμε για 47,7 δις ευρώ κάποιος ευρωβουλευτής είπε εντάξει τώρα τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έρχονται στην Κροατία κατά τη διάρκεια της προενταξιακής διαδικασίας και τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά που σας λέω, που φύγαν από τη χώρα. Δημόσιο χρήμα είναι αυτό. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. μπορεί να ασκήσει κάποιο είδου κοινοβουλευτική πίεση στην Κροατία ώστε να διερευνήσει αυτά τα σκάνδαλα, ώστε να επιστρέψουν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα χρήματα στη χώρα. Κάποια από αυτά σίγουρα μπορούν να, να, να ε, επιστραφούν, γιατί ξέρουμε που βρίσκονται, στις εταιρείες, σε ιδιώτες, σε ε, ε, ε, δραστηριότητες εξαγοράς κινήτων. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα μπορούν να επιστραφούν στην Κροατία και είναι πολύ περισσότερα από όσα θα πάρει η Κροατία από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αν με ρωτάτε, υπάρχει, μάλλον υπάρχει εγγύηση ότι θα χρησιμοποιούν σωστά αυτά τα χρήματα τα ευρωπαϊκά. Όχι, δεν υπάρχει εγγύηση. Γιατί δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου ξεκάθαρη η διαφάνεια στη χρήση αυτών των κονδυλίων. Άμα έρθετε στην Κροατία και ρωτήσετε τι κάνετε, έχετε διαφανείς διαδικασίες για να απορροφήσετε αυτά τα κονδύλια. Βέβαια, θα σας δώσουν ένα σωρό εκθέσεις, ότι όλα γίνονται με διαφάνεια, ότι όλα γίνονται νομίμως, ότι όλα δημοσιεύονται κτλ. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που καταχράστηκαν τα κροατικά χρήματα είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστούν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Και δεν υπάρχει, δεν ασκείται καμία πίεση για να γίνουν όλα αυτά να νομιμοποιηθούν και να υπάρξει διαφάνεια. Εδώ σίγουρα μπορείτε να βοηθήσετε, να ασκήσετε πίεση σε αυτούς. Και όπως είπα και νωρίτερα, ως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε επίσης να μας βοηθήσετε να ασκήσετε πίεση στην Κροατία ώστε αυτή η νομοθεσία για την προστασία των ανθρώπων που μιλούν για τη διαφορά, να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, να έρθετε στην Κροατία, να πιέσετε ώστε να υπάρξει νομοθεσία για την προστασία των ε, δημοσιογράφων έρευνα, γιατί διαφορετικά θα επικρατήσει άκρα σιωπή στην ε, Κροατία. Ευχαριστούμε κύριε Μάρκετ. Καλό το συναδέλφους να το σκεφτούν <laughs> όλα αυτά. Η Κροατία από την 1η Ιουλίου θα γίνει μέλος της Ένωσης. Και τα όσα μόλις ακούσαμε είναι σοβαρότατες καταγγελίες, κατηγορίες. Ανήκουστα πράγματα. και δεν διαφέρουν και πολύ από πραγματικότητες που ήδη ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτη-μέλη και μάλιστα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ένωσης. Παρακαλώ πρώτο ερώτημα για το τραπεζικό απόρριτο. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να κινηθούν σωστά και με ένα ευρώ θα παίρναμε το αντίτιμο, δηλαδή ένα αγαθό αντιστοιχίας που να στοιχίζει ένα ευρώ, όχι να έχουμε 5 προς 1. Γι' αυτό, αν μειωθεί το τραπεζικό απόρριτο, αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα. Πολλά προβλήματα δεν θα υφίσταντο. Το δεύτερο ερώτημα. Πόσες εκθέσεις οδηγούν σε δίωξη. Έχουμε αριθμητικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Έχουμε τις καταδίκες. Μπορείτε να δείτε τα ποσά και βλέπετε ότι μόνο πέντε χώρες προέχουν, Ηνωμένο Βασίλειο χίλιες καταδίκες, 500 στην Ολλανδία, 400, ε, Δανία πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση με το πληθυσμό, διότι το δανέζικο σύστημα καθιστά πιο εύκολο για τον εισαγγελέα να κάνει δίωξη για ε, ξέπλυμα, ενώ στις άλλες χώρες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Δανία είναι πολύ αποδοτική, η άλλη λιγότερο. Η Γερμανία βρίσκεται στο μέσον. Στην Ολλανδία έχουμε ένα, να κάνουμε με ένα 0,5% που οδηγεί σε καταδίκη με βάση τον αριθμό που σας είπα, τους 400 δηλαδή. Ε, το γεγονός, ε, η αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ε, καταγγελιών και καταδικών δεν υπάρχει, καταδίκης δεν υπάρχει. Προτείνω στην Επιτροπή τα εξής. Πρώτον, η τρίτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ξεπλήματος μας οδήγησε σε πολύ μικρές αλλαγές, αλλά προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι η τέταρτη οδηγία θα ενέχει τα ίδια. Τώρα, ως προς τη φοροδιαφυγή, άλλαξα γνώμη μετά από τις διαρροές. Θεωρώ ότι πρέπει να διώκεται με άλλους τρόπους από κοινωνικά κινήματα ή μέσα, άρα να μην ενταχθεί στην οδηγία. Θα ήθελα όμως να ε, ξέρετε από τα κράτη-μέλη τι σημαίνει ε, φορολογικό έγκλημα στα 27 κράτη, γιατί είμαι σίγουρη ότι σημαίνει διαφορετικά πράγματα στις χώρες. Να έχετε συνολική εικόνα λοιπόν για τα τι περιλαμβάνει το φορολογικό έγκλημα. Προστατεύστε επίσης τα κράτη-μέλη. Έχουμε συγκρουόμενες ρυθμίσεις και πολλές φορές τα, ε, ε, τα σχέδια της ΦΑΤΦ δεν είναι ίδια για όλους. Δηλαδή, τι πρέπει, πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε αμοιβαία τις ε, τραπεζές μας. Δηλαδή, η οδηγία λέει ναι, μπορούμε να εμπιστευτούμε, αλλά αν δεν πληρούνται τα πρότυπα και οι προδιαγραφές της ΦΑΤΦ, τότε δεν φτάνουμε πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν να είσαστε πιο επιθετικοί, δηλαδή υπάρχει νόμος για τα κράτη-μέλη, δεν μπορείτε να έχετε ένα διαφορετικό, ένα διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεσπόζει δηλαδή το κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει να είναι παγκόσμιος παίκτη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερο από ό,τι ισχύει τώρα, με βάση τα πρότυπα, τα πρότυπα της ε, ΦΑΤΦ. Και χρησιμοποιήστε τη φοροδιαφυγή έτσι ώστε να γίνεται πιο διαφανής. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έξω από αυτές τις ε, αποφάσεις χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Με τη φοροδιαφυγή μπορεί να ενταχθεί και το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία μέσω ανοιχτής συζήτησης γιατί βρισκόμαστε σε μία μεταδημοκρατία και οι χρηματοπιστωτικές αγορές ορίζουν τον κοινοβουλευτισμό. Θα πρέπει να ισχύσει όμως το αντίθετο. Τώρα, ποιες ώρες ε, δεν καλύπτονται από τη ΦΑΤΦ. Θα πρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε την Αγγόλα, την Αιθιοπία, το Ιράν και τη ε, Νότια και την Βόρεια, με συγχωρείτε, Κορέα. Υπάρχει ο μαύρος κατάλογος, αλλά το ζήτημα είναι τι επιπτώσεις έχει. Γιατί μπορεί να υπάρχει δίθεν συμμόρφωση, ιονή συμμόρφωση, δηλαδή διαδικασία copy-paste, αλλά στην ουσία δεν ε, γίνεται, δεν υπάρχει ίδια μεταχείριση. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινό παρονομαστής. Οι χώρες έχουν ε, πολλές δυνατότητες να βρουν παραθυράκια. Δεν πρέπει να έχουμε μία διτή συμμόρφωση. Τώρα το ότι κατονομάζουμε και ξεμπροστιάζουμε νομίζω ότι, θα πρέπει να γίνει, ότι δεν θα πρέπει να γίνει. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό το ξεμπρόστιασμα των ε, χωρών. Αυτό λειτουργεί στις ε, επιχειρήσεις, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όχι όταν μιλάμε για τον δημόσιο τομέα που βασίζεται στους μεγάλους ε, δωρητές. Το naming and shaming μπορεί να ισχύσει σε, για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ε, οι επιχειρήσεις, δηλαδή για το Starbucks που το κοινό δεν αγοράζει τα προϊόντα του, αλλά όταν μιλάμε για την Κύπρο αυτό δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό, όχι μέσω επισήμων οργανώσεων. Επίσης εμπιστεύομαι τα κοινωνικά κινήματα. Πολλοί ε, δεν είναι ευχαριστημένοι και οι διαρροές ε, θα έχουν μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για κινήματα όπως το ΑΤΑΚ και άλλα. Ε, στατιστικά στοιχεία δεν τα χρειαζόμαστε ευπρόσδεκτα βεβαίως. Η Eurostat και η σχετική γενική διεύθυνση έχουν ασχοληθεί, αλλά η κατάρτιση τους είναι χρονοβόρα. Δεν πρέπει να πάρουμε τις πρώτες ε, διώξεις και καταδίκες και να πούμε «Α, η Ολλανδία είναι στο 3, η άλλη χώρα είναι στο 1. Οι στατιστικές είναι χρονοφόρες, ιδιαίτερα ως προς τις εκροές. Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε, ας βασιστούμε στο input, δηλαδή πόσο δαπανούν οι χώρες για το ξέπλυμα, ε, τι πληροφορίες υπάρχουν Ας μετρήσουμε τις προσπάθειες, διότι τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Για την ανεργία, ας πούμε, ήταν διαφορετικές οι μετρήσεις, με βάση διαφορετικές μεταβλητές. Τώρα ε, υπάρχει κοινό πρότυπο για να μετρήσουμε την ανεργία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει με, κοινούς συντελεσ... ε, με κοινές μεταβλητές, με για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τυχαία αριθμητικά στοιχεία και να τα συγκρίνουμε. Στη Γερμανία ο σπονδιακός χαρακτήρας ε, υπερισχύει. Δηλαδή τα κρατήδια είναι υπεύθυνα για την φοροδιαφυγή και ε, δυστυχώς μερικά κρατήδια είναι πιο αυστηρά από άλλα. Ο ομοσπονδιακός λοιπόν αυτός χαρακτήρας είναι δύσκολος. Η Γερμανία έχει προβλήματα αλλά δεν θέλω να μπω σε τέτοια θέματα. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή βεβαίως, αλλά έχει σημασία ποιο πρότυπο θα ακολουθήσουμε. Πολλά συζητώνται και οι δημόσια εισαγγελία είναι διαφορετική. Από χώρα σε χώρα άλλοι συνδράμονται από τις αστυνομικές αρχές, υπάρχει διακριτική ευχέρεια. Άλλες εισαγγελικέ αρχές πρέπει να συνδιαλογούν με το δικαστή πριν αρχίσουν τη δίωξη. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικά ιστορικά συστήματα. Γι' αυτό και η επιλογή θα ορίσει κατά πόσο θα έχουμε ένα σύστημα που θα δεσπόζει ή όχι. Τέλος. Είπατε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε το ξέπλυμα. Εγώ έχω αφιερώσει μια ζωή σε αυτό. Μόνο το σκληρό έγκλημα ε, έχει κατατροποθεί, αλλά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπορεί να μετρηθεί από διαφορετική οπτική γωνία και φτάνουμε σε ένα τρίγωνο, σε έναν τριγωνισμό με βάση τις διαφορετικές ε, οπτικές γωνίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε ένα μέσο όρο. Μιλάμε για 2 με 5% του ΑΕΠ. Αυτά είναι τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, προβαίνουμε σε εικασίες και έχουμε εκτιμήσεις, οι οποίες βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα. Έχουμε και ένα ε, ιταλικό μοντέλο από έναν ε, φορέα στη Ρώμη που κάνει συνεχείς μετρήσεις ξεπλήματος. Και σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, στις ΙΠΑ αυξάνεται το ξέπλυμα, ενώ στην Ευρώπη ακολουθεί φθήνουσα πορεία. μερικό τουλάχιστον. Άρα τα ναι. μέσα που χρησιμοποίησαμε ήταν κάπως αποδοτικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη παρέμβαση την κυρία Σπαπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Έχω ακούσει δύο-τρεις φορές την αναφορά στην Κύπρο. Είμαι Κύπρια ευρωβουλευτή. Δυστυχώ ήθελα να έρθω πιο ενωρί, αλλά οι πτήσει από την Κύπρο είναι δύσκολε. Ταξιδεύω από τι 3 το πρωί για να φτάσω τώρα γιατί αλλάζουμε δύο πτήσει. Ε, έχω ακούσει ότι η τελευταία μιλήτρια έχει αναφερθεί στην Κύπρο και μάλιστα είπε ότι δεν είναι στον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων και ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό το money laundering και επίσης το tax evasion ότι είναι problem of the rich countries. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που λέτε. Όμω, εγώ είμαι Ευρωβουλευτή από το 2009 και έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, λίγο πριν από το haircut, πολλέ άδικε και τεκμηρίωτε ε, κακόπιστε επιθέσει εναντίον τη χώρα μου. Άκουσα από Τσέχο συνάδελφο και από Γερμανό συνάδελφο και από Σουηδό να λέω ότι η Κύπρος είναι τάχα χώρος ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και παράνομων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Θα πω απλά ότι παρακολουθώ το θέμα γιατί ήμουν για 9 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εκπροσωπώντας το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και θα σας δώσω και links, μπορώ να τα στείλω σε όλους τους ενδιαφερόμενους. το Manival, που είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάνει έλεγχο και υπάρχει έκθεση 27 Σεπτεμβρίου 2011. Ο τίτλος είναι στα γαλλικά, θα σας το στείλω αν θέλετε και λέει ακριβώς ότι δεν επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία λέγονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε και εφαρμόζει πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και επίσης υπάρχει και από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και μάλιστα πρόσφατο, 5 Μαρτίου 2013, υπάρχει μια συγκριτική μελέτη που ονομάζεται Money Laundering and Financial Crimes και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος πληρεί όλα τα κριτήρια καταπολέμησης του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος σε όλες τις κατηγορίες μέτρων και μιλούμε για 20 κατηγορίες. Ενώ αντίθετα αυτοί που κατηγορούν την Κύπρο για να δικαιολογήσουν το άδικο haircut το οποίο επιβλήθηκε στη χώρα μου, το οποίο ήταν εκατάστρεψε το οικονομικό μοντέλο και κατάστρεψε την οικονομία και τον λαό και θα χρειαστεί κόπος και χρόνια για να επανακτήσουμε ακριβώς το σθένος μας και την οικονομία. Δυστυχώς εδώ υπάρχει αναφορά ότι η Γερμανία, η Σουηδία και η Τσεχία παρουσιάζουν κενά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες μέτρων και αυτό υπάρχει πάνω στην ιστοσελίδα. Καταλήγω θεωρώ πολύ άδικο και ανέντιμο. I finish, I finish. Εγώ συμφωνώ να αρθεί το τραπεζικό απόρριτο. Το πρόβλημα της Κύπρου ήταν η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στο κούρεμα που αποφάσισε το Eurogroup των χρεών των ελληνικών τραπεζών που στήχησε στη χώρα μου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ που σημαίνει 25% του ΑΕΠ. Επομένω, αν ζητήσαμε βοήθεια 5,8 δι, είναι γιατί τα 4,5 ήταν το κόστο που πλήρωσε η Κύπρος από ακόμα μια λαθασμένη απόφαση για τον τρόπο που απέτυχε το Eurogroup να εφαρμόσει το κούρεμα χρέου στην Ελλάδα. Και τελειώνω, νομίζω ότι είναι λάθο να γίνεται αναφορά στην Κύπρο. Εγώ μπορώ να αναφέρω πολλού φορολογικού παραδείσου. Είναι το Isle of Man, είναι το Σαν Μαρίνο, είναι το Γιβραλτάρ, και πολλέ άλλε χώρε. Αν χαμηλούμε για την Κύπρο, έχουμε πολλά να πούμε για πολλέ άλλε χώρε και είναι λάθο να γίνεται αυτή η αναφορά. Σα ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Όχι, δεν μιλήσαμε στην πράξη για την Κύπρο. Μιλήσαμε για διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που ήταν το σημαντικό ήταν οι προδιαγραφές διαφάνειας, οι οποίες θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν ακριβώς για να αποφεύγουμε προβλήματα τέτοιου τύπου. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας και <coughs> τους εισηγητές μας για τις ομιλίες τους και κυρίως για τα σημαντικότατα νέα που μας έδωσαν κήρυσω το πέρα της και θα ξαναρχίσουμε στις 3 ε, ε, στην ίδια αίθουσα.